Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Uh, Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αυτή τη δεύτερη μέρα συνεδριάσεων της Επιτροπής μας. Και το σημερινό είναι πρόγραμμα ιδιαίτερο, μια ομάδα εργασίας με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Από κοινού με την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας υπό την αιγίδα βεβαίως και την καθοδήγηση της ε, υπηρεσίας πολιτικής. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή συνεδρίαση. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου κύριος Ηλίου Βίγκλας, είναι και εδώ, είναι εδώ επίσης. Πρώτη φορά έχουμε τέτοιου είδους συνεδρίες, αλλά η Πολωνία και η Ρουμανία έχουν ε, μάθει να συνδυάζουν τις δυνάμεις τους. Και επίσης μπορούμε να έχουμε την παρουσία των εμπειρογνωμόνων μας που πρόκειται για εργαστήριο. Δίνω το λόγο μέσα στον κύριο Ηλίου Βίνκλερ και μετά θα κάνουμε την ε, παρουσίαση των διακεκριμένων ειδικών μας. Κύριε Βίγκλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, διακεκριμένοι, προσκεκλημένοι, διαφόρων θεσμικών οργάνων, βιομηχανίας με κυβερνητικών οργανώσεων, και βέβαια οι εγκριτοί ομιλητέ που είστε εδώ για να μιλήσετε για το θέλαμα αυτό. Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Επιτροπής Εθνούς Εμπορίου. Αντιπρόεδρος μόνο συμμετέχει στην εκδήλωση αυτή. Μιλούσα για τον πρόεδρο, δεν ξέρω αν ε, αυτό είναι ο λόγο που δυνάμωσε ξαφνικά το μικρόφωνο. Ο κύριο Λάγκεν, λοιπόν, πρόεδρο τη Επιτροπή μα, ε, δεν μπόρεσε να είναι παρόν σήμερα. Έτσι εκπροσωπώ εγώ την ΙΝΤΑ, Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Και γι' αυτό σας καλώ να συστήσουμε ένα θέμα πολύ σημαντικό Πρέπει να γίνει μια ουσιαστική και καλή μεταρρύθμιση του πλαισίου, νομοθετικού πλαισίου για τα προϊόντα διπλής χρήσης. Και νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο μερίδιο του, της ομοφανίας που αφορά αυτός ο τομέας Άρα πρέπει να γίνει μια σωστή ανάλυση και επιλογές πολιτικές. Γιατί έχουμε να κάνουμε με χιλιάδες μικρές και μεσές επιχειρήσεις με θέσεις εργασίας υψηλού ή προσθέμενης αξίας που αποτελούν τη ράχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η υλοποίηση αποτελουν τη κοκαλια της νομοθεσίας θα ε, αφορά στη συνέχεια τις εθνικές αρχές. Επίσης έχουμε να κάνουμε με έναν μηχανισμό πολύ σοβαρό και στεναρό, μηχανισμό ελέγχου δηλαδή που θα χρειαστεί, για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, για να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια έκφραση από την αλληλεία πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να πιάνουμε τους μεγαλοκαρχαρίες, αλλά να μην κάνουμε ζημιά στη Μαρίδα. Και επίσης, για να πω κάτι άλλο πολύ πιο καθημερινό, αν μου επιτρέπει ο Πρόεδρος, δεν πρέπει μαζί με τα ξερά να καίμε και τα χλωρά. Αυτές είναι οι ευαισθησίες που έχουμε, στις αποφάσεις που έχουμε να λάβουμε. Πρέπει να γίνονται ε, επικαιροποίηση των παραρτημάτων με την κατεξουσιοδότηση διαδικασία και, να... και αυτό ισχύει μέχρι τώρα. Πρέπει να γίνει ο μηχανισμός πιο αποτελεσματικός και έγκαιρος στην αντίδρασή του. Πρέπει να σταθούμε σε μια κοινοτική προσέγγιση, να εναρμονιστεί περαιτέρω το σύστημα για να αποτραπούν οι στρεβλώσεις, οι διαφορές, και τα προβλήματα σε σχέση με τον ε, έλεγχο των εξαγωγών προϊόντων τρίτης χρήσης και επίσης χρειάζεται συνεργασία των κρατών μελών για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Δεν θα σας καθυστερήσω άλλο πρόεδρε και σταματώ. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Winkler. Now... Ευχαριστώ κύριε Βίνκλερ. Επιτρέψτε μου τώρα να παρουσιάσω τον πρώτο ομιλητή εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, τον κύριο Πάολο Γκαρτζότη. Ελπίζω να, προσφέρω, να προφέρω καλά το όνομά σας. Ο κύριος Πάολο Γκαρτζότη είναι τμήματάρχης ε, του τμήματος που είναι υπεύθυνο για τα προϊόντα διπλής χρήσης και θα ήθελα να σας ζητήσω στην αρχή της παρουσίασής σας να μας πείτε δύο λόγια για την ε, αρμοδιότητα και την εντολή του τμήματός σας. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Ιαν Στιούαρτ, ο οποίος ε, είναι από το King's College του Λονδίνου, επικεφαλής του, τμήμα, του προγράμματος Α, που ασχολείται και πάλι με τους ελέγχους των προϊόντων διπλής ε, χρήσης και τη δόκτωρα Σίμπιλ Μπάουερ από το ΣΥΠΡΙ, ε, την πρωτοβουλία της Στοκχόλμης δηλαδή. Χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση, θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο απευθείας στους εμπειρογνωμονές μας, ξεκινώντας με τον κύριο Γκαρτζότη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Όπως είπε η Πρόεδρος, είμαι επικεφαλής του τμήματος που ασχολείται με τα ε, προϊόντα διπλής χρήσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια μικρή καλή ομάδα που ασχολείται με τα θέματα αυτά και είναι όλοι εδώ στην αίθουσα. Ο Στεφάν Σαντών, ο Μάριο Ασκολέζε και καθήκον μας είναι να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την αναθεώρηση των ελέγχων των εξαγωγών όπως ζητήθηκε από τους νομοθέτες, από εσά δηλαδή, βάσει του άρθρου 25 του κανονισμού. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στην πρώτη διαφάνεια γιατί δεν ξέρω πώς θα τη γυρίσω. η έλεγχη των εξαγωγών δεν ήταν αναγνωρισμένη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ε, εκεί είχαμε μια πρώτη απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ξεκίνησε λοιπόν ε, η εκπόνηση κοινών κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι τελικά ήταν απλώς μια κωδικοποίηση του ελάχιστου κοινού παρονομαστή, αυτών ε, τον οποίο ε, τα οποία εφαρμόζονται στην εθνική νομοθεσία. Η ιδιομορφία του τομέα είναι ότι Υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του άρθρου 207 για το εμπόριο. Είμαστε λοιπόν αρμόδιοι για να προτείνουμε νομοθεσία αλλά αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει το ζήτημα αυτό και ασχολούνται με την έκδοση αδειών για εξαγωγές είναι τα κράτη-μέλη που ε, είναι αρμόδια για τις εξαγωγές αυτές. Για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία για να μπορούμε να έχουμε και αυτή την εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών. Είχαμε ένα πρώτο κανονισμό λοιπόν το 2000, ε, μετά από τις απειλές ε, στην αρχή του αιώνα για τρομοκρατικές επιθέσεις είχαμε μια κρίσιμη στιγμή, εκεί εγκρίθηκε και μια νέα στρατηγική για την διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής το 2003 και σιγά σιγά φτάσαμε στην ε, δεύτερη αναδιατύπωση του κανονισμού για τα προϊόντα διπλής χρήσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο κανονισμός ο οποίος είναι ενισχύει αυτή τη στιγμή του 2009. Ο κανονισμός αυτός ήδη ζητούσε μεταρρύθμιση και βελτιώσεις και στόχο είχε να επιτύχει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μας ε, του κλάδου και των εξαγωγέων και της ασφάλειας, όπως έλεγε και ο τίτλος. Ξεκινήσαμε ε, το 2011 ένα διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση μια πράσινη βίβλο και αυτό οδήγησε τελικώς ε, στα ουσιαστικά στοιχεία των προτάσεών μας και των ιδεών μας και θα ήθελα να καλέσω όσους ασχολούνται με το θέμα αυτό να δουν την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014 όπου υπάρχουν κάποιες ιδέες τις οποίες θα σας παρουσιάσω εντάχει σήμερα και έχουν συμπεριληφθεί εκεί. Από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι μια πολιτική δήλωση μέχρι την ουσιαστική πρόταση κανονισμού Χρειάζεται, όπως γνωρίζετε, και εδώ ίσως μπορούμε να περάσουμε και στην επόμενη διαφάνεια, ε, χρειαζόμαστε μια αξιολόγηση επιπτώσεων. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες ε, που περιλαμβάνονται σε αυτή τη διαφάνεια, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τουλάχιστον στη βάση. Ε, δεν είναι εύκολο να ορίσουμε τον όλο κλάδο προϊόντων διπλής χρήσης, διότι οποιοδήποτε τομέος μπορεί ε, να θεωρηθεί ότι ε, ασχολείται με εξαγωγές ε, προϊόντων διπλής χρήσης. Επομένω, προκειμένου να διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι μας, έχουμε μια πρώτη διαδικασία. Από εκεί και πέρα θα περάσουμε στην ανάλυση των δεδομένων και βάσει της ανάλυσης των δεδομένων θα δούμε τι επιλογές θα μπορούσαμε να προτείνουμε στο τελικό σχέδιο έκθεσης. Θα έχουμε και μια δημόσια διαβίλευση. θα δούμε λοιπόν ε, ε, και τα αποτελέσματά της, θα δημοσιευτούν ε, τον Ιούλιο κατά πάσα πιθανότητα. Το καλοκαίρι λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε στην παραλία, μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Και φυσικά για την αξιολόγηση επιπτώσεων να σας πω ότι επαφίεται στην εμπειρογνωμοσύνη του Σύπρη πρωτίστως και θα ακούσουμε αργότερα τον εκπρόσωπο του Σύπρη ε, διότι έχουν μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη ε, επί του ζητήματος. Τώρα, γιατί θέλουμε να αναθεωρήσουμε και να βελτιώσουμε τους ελέγχους των εξαγωγών. Καταρχάς, όσον αφορά ε, την ασφάλεια, ε, το περιβάλλον ασφάλειας έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Θα θέλαμε να επικεντρωθούμε σε κάποια σημεία. Όταν ε, δημιουργήθηκαν οι έλεγχοι των εξαγωγών, ε, ήταν πολύ απλουστευμένοι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν τεχνολογία που ε, ήθελαν να μην πέσει στα χέρια άλλων κρατών που δεν μοιράζονται τις ίδιες αξίες. Αυτά έχουν αλλάξει πλέον και πλέον υπάρχουν διεθνείς ε, απειλές ασφαλείας. Αν δει κάποιος τις ειδήσει τη σήμερα ημέρα το καταλαβαίνει αμέσως και φυσικά είναι αυξημένες οι απειλές από μη κρατικούς φορείς και όταν αναφέρουμε σε μη κρατικούς φορείς ε, δεν αναφέρομαι μόνο στο Ισλαμικό κράτος, στο ISIS αλλά μπορεί να υπάρχει και κάποιος ε, ανύποπτος ε, μάλλον, άνθρωπος υπεράνω υποψίας ο οποίος ε, μπορεί να παρισφρήσει στην ε, αλυσίδα διανομής και να αποτελεί κίνδυνο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ε, βεβαίως υπάρχουν και παραδοσιακά κρατικά προβλήματα, παραδείγματος χάρη προβλήματα με τη Βόρεια Κορέα, Κορέα ή τη Συρία. Επίσης έχει αλλάξει το επιστημονικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Πριν από 20 χρόνια, προκειμένου κάποιος να διακινήσει αγαθά, έπρεπε να ε, υπάρχει ε, μια συσκευή, να περάσει κάποιος τα σύνορα και να την παραδώσει σε κάποιον. Σήμερα έχει αλλάξει το περιβάλλον ασφαλείας, υπάρχει βέβαια σαφώς το θέμα της κυβερνοασφάλειας, οι απειλές μέσω διαδικτύου είναι πάμπολες, αλλά επίσης υπάρχει και το cloud computing, υπάρχει δυνατότητα δηλαδή μεταφοράς τεχνολογίας με άλλο τρόπο ε, και στο μέλλον θα υπάρχει και δυνατότητα, για παράδειγμα, τρισδιάστατης εκτύπωσης αγαθών. Είναι σαφές λοιπόν ότι ε, είναι πολύ πιο προηγμένες οι απειλές από αυτές που είχαμε στο παρελθόν. Φανταστείτε επίσης ζητήματα όπως η επιστημονική έρευνα. Η επιστημονική έρευνα ε, είναι εξαιρετικά προηγμένη και μπορεί να ε, αποτελέσει πολύ σημαντική πρόοδο προς όφελος της κοινωνίας, αλλά μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί και την επιστημονική έρευνα για την ε, μετάδοση ευαίσθητων ε, δεδομένων. Υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για μια έρευνα για βιολογικά δεδομένα για εμβόλιο κατά της γρήπης και εκεί υπήρξαν και κάποιες νομικές συνέπειες σε κάποιο κράτος μέλος, διότι η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε σε ξένα έντυπα χωρίς να υπάρχει απαραίτητη άδεια. Και το τελευταίο σημείο που έχουμε εδώ στη διαφάνεια αυτά είναι το οικονομικό περιβάλλον. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε μορφή εμπορίου. Δεν παράγονται απλώ αγαθά και εξάγονται σε, μια χώρα και εξάγονται σε μια άλλη. Λειτουργεί τελείω διαφορετικά ο κόσμο σήμερα ο καθής συνεισφέρει ένα λιθαράκι στην αλυσίδα διαμονής. Οι περισσότεροι από εσά, για παράδειγμα, έχετε ένα τηλέφωνο στην τσέπη σας. Αν προσπαθήσετε να εξηγήσετε ποιος ε, είναι υπεύθυνο για την εξαγωγή του τηλεφώνου, δεν είναι σαφές. Επομένως, η έλεγχη για τα προϊόντα διπλής χρήσης και το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, και από πλευράς ε, ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας. Επίσης είναι θολά τα όρια μεταξύ ε, στρατιωτικής και πολιτικής βιομηχανίας. Ε, αυτό ήταν σαφές στο παρελθόν, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές καινοτομίες και τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως ε, για τον ένα ή για τον άλλο σκοπό και για πολιτικούς και για στρατιωτικούς σκοπούς. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε στρέβλωση στους ελέγχους στρέβλωση του εμπορίου και θα μπορούσε αυτό να υποσκάψει και την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγέων μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Αν υπάρχει ε, στρέβλωση του ανταγωνισμού, τότε δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η ασφάλεια πλήττεται, διότι αν έχουμε διαφορετικούς ελέγχους σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε υπάρχει δυνατότητα άγρας του κατάλληλου χώρου για αυτούς που δεν χρησιμοποιούν ε, για καλό σκοπό το σύστημα. Έχουμε λοιπόν διάφορες πραγματικότητε που παρουσιάζονται σε αυτή τη διαφάνεια, τη έχουμε βάλει σε διάφορα πλαίσια. Καταρχάς πρέπει να προσαρμοστούμε στο περιβάλλον ασφαλείας που εξελίσσεται συνεχώ, δεύτερον να προωθήσουμε ισότιμους όρου ανταγωνισμού, τρίτον να αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό καθεστώ ελέγχου των εξαγωγών και να έχουμε ε, αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή. Να περάσω τώρα ε, στο πρώτο σκέλος που είναι η προσαρμογή σε αυτό το περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, υπήρξε πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά η σχέση μεταξύ ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταρχάς. Ε, εμείς αυτό το αποκαλούμε ανθρώπινη ασφάλεια, αλλά αυτό είναι ένας τίτλος όπως κάθε άλλον. σήμερα πρέπει να περάσουμε πέραν της έννοιας της ασφάλειας του κράτους και εσωτερική-εξωτερική ασφάλεια. Πρέπει να λάβουμε υπόψη στους ορισμούς που χρησιμοποιούμε την ασφάλεια των ατόμων, την ασφάλεια των λαών, την ασφάλεια που σχετίζεται με την τρομοκρατία. Κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και να αλλάξουμε τα κριτήρια ελέγχου, όπως έχουμε και πει και προηγουμένως, ώστε να μπορέσουμε να προβλέψουμε κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε όλο ένα και περισσότερο υπόψη της απειλής μέσω κοινωνίας της πληροφορίας και επικοινωνίας. Πολύ πρόσφατα, λόγω των παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων που ξεκίνησαν με τεχνολογίες οι οποίες αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε σημαντικές απειλές κατά προσώπων και αυτή τη στιγμή ε, έχουμε καταφέρει με ένα από τα καθεστώτα που καθορίζει ε, τα προϊόντα τα οποία ελέγχονται να περιορίσουμε τη χρήση αυτών των τεχνολογιών για αυτούς τους σκοπούς. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι αυτή η ευφυής ασφάλεια, δηλαδή η δυνατότητα να ανταποκρίνεται κάποιος ταχύτατα στις αλλαγές ε, λόγω των τεχνολογικών προκλήσεων. Και εδώ, κατ' ουσίαν, έχουμε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα υπάρχει απλώς μία αρχή που θα είναι υπεύθυνη για την αδειοδότηση, ένας κρατικός έλεγχος και το καθεξής. Δεν αρκούν αυτά, πρέπει να υπάρχει ατομικός έλεγχος στα σύνορα, θα πρέπει να δίνονται κατευθυντήριες γραμμές στους εξαγωγείς για να διευκρινίζουν κάποια πράγματα για τις τεχνολογίες. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε και εμείς τη συνεισφορά μας ε, στα διάφορα ζητήματα. Τέλος, όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των ελέγχων, αλλάζει ο κόσμος, επομένως πρέπει να αλλάξουμε και εμείς κάποιους από τους ορισμούς που έχουμε τι είναι ένας ε, προμηθευτής με τις αλλαγές που έχουμε στα παγκόσμια συστήματα και με τις διαφορετικούς φορείς ε, που συμμετέχουν στην αλυσίδα διανομής είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το εξετάσουμε στην αναθεώρησή μας. Επίσης, το θέμα της δικαιοδοσίας. Ε, δεν θέλουμε να πάμε ε, μέχρι του σημείου που πάνε οι Αμερικανοί που έχουν και εφαρμογή εκτός Ηνωμένων Πολιτειών αλλά εάν κάποιος δραστηριοποιείται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, συμμετέχει ενεργά στη διακίνηση αγαθών διπλής χρήσης για κακόβουλο σκοπό, τότε πρέπει κάπως αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Και τέλος, για να μην μακρηγορήσω άλλο, Υπάρχει αυτή η άειλη μεταφορά γνώσης που ανέφερα και προηγουμένως, η ITT, η επιστημονική έρευνα και η μεταφορά αγαθών που δεν είναι υλικά αγαθά, κάτι το οποίο γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικό σήμερα. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι προηγουμένως σταθήκαμε στις πτυχές ασφαλείας, εδώ έχουμε τα οικονομικά στοιχεία, την ανταγωνιστικότητα κλπ. Πώς λοιπόν θα βοηθήσουμε ώστε να βοηθήσουμε τις εταιρείε μας με συνθήκες ασφαλείας. Έχετε καταρχάς ε, την επικυριοποίηση του πίνακα των ε, παραρτημάτων όπου έχουμε τα κατάλογο των αγαθών πρώτα απ' όλα το πιο σημαντικό και έπρεπε να, περάσουμε, να περάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ε, τακτική νομοθετική διαδικασία για να το καταφέρει αυτό. δεδομένου και του κατεπίδοντος βέβαια δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε ένα-δύο χρόνια μέχρι να επικαιροποιείται ο πίνακα κάθε φορά και γι' αυτό έχουμε προτείνει τώρα την κατεξουσιοδότηση διαδικασία ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να προχωρούμε πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά και με πιο προηγμένο τρόπο στο μέλλον. Αυτό που έχουμε υπόψη λοιπόν στις ιδέες μας ενώπιση του κανονισμού, του νέου κανονισμού, είναι να εξεταστεί μια νέα σειρά, νέοι τύποι αδειών. Δηλαδή να ξεφύγουμε από την ιδέα ότι χορηγείται μία άδεια για κάθε συναλλαγή, η παραδοσιακή διαχείριση δηλαδή, και να κοιτάξουμε ένα σύστημα ανοιχτό αδειοδότησης, όπου περισσότερες της μίας αδείες θα μπορούσαν να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα συναλλαγών και δι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε περισσότερο ε, γενικευμένο ευρωπαϊκό σύστημα αδειοδότηση εξαγωγών ορισμένων αγαθών προ ορισμένε κατευθύνσεις που θεωρούνται, στους ορισμένου προορισμούς που θεωρούνται επαρκώς ασφαλείς επί παραδείγματι. Άρα χτύνουζουμε θα έλεγα έναν ψηλότερο τοίχο αλλά γύρω από ένα μικρότερο κήπο. Σε αυτές τις διευκολύνσεις θα μπορούσαν να εντάσσονται αποστολές χαμηλότερης αξίας, διακοινωτικές ε, μεταβιβάσεις τεχνολογίας, μάλλον δια, διαεπιχειρησιακές, εντός του ίδιου ομίλου δηλαδή, ο έλεγχος του πυρηνικού υλικού μπορεί να καλυφθεί από το τροποποίηση του πρωτοκόλλου παριθμών 4, Και αντίστοιχα παρακολουθούμε τις συνθήκες που επικρατούν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σε σχέση με το Βιετνάμ έχουν απέτηση 500 ε, κιλών για την άδεια. Αυτά λοιπόν κοιτούμε να κάνουμε και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί και η παγκόσμια σύγκληση. Ε, βεβαίως για να εξασφαλιστεί αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε στις διάφορες ρυθμίσεις. η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία από τις διαπραγματεύσεις είναι παρατηρητής μόνο, σε άλλες δύο ως Ένωση, αλλά μόνο εάν τα κράτη-μέλη προσετεριστούν ή ενστεριστούν αυτές τις ρυθμίσεις μπορεί να καταστούν ευρωπαϊκές. Ε, για να κλείνω γιατί βλέπω ότι έχω μακρηγορήσει. Στην επόμενη διαφάνεια για το πώς μπορούμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα εξαγωγών και ανταγωνιστικό ταυτόχρονα. Αυτό που ήθελα εγώ να σημειώσω είναι ότι δεν χρειάζεται πάντα να ρυθμίζονται ε, από την νομοθεσία, γιατί πολλά μπορούν να εξακαλυφθούν από το ήπιο δίκαιο, από τις κατευθυντήριες γραμμές, η εναρμόνιση παραδείγματι. Ε, ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, παραδείγματι. Αυτό έχει ήδη εξασφαλιστεί και στα τελωνία, στο εμπόριο και μπορούμε νομίζω να το επιτύχουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα προϊόντα διπλής χρήσης. Ένα ζήτημα ιδιαίτερη σημασία είναι η συλλήβδην έλεγχη, το catch-all όπως λέγεται, ε, παράδοξο όνομα κάπως, αλλά αφορούν αυτή η στοιχεία για τα οποία έχουμε πληροφορίες πως χρειάζεται να επιλευθευθούν και εκεί όταν υπάρχει λόγος, ε, λόγος ασφάλειας ή ανταγωνιστικότητας πρέπει να παρακολουθούμε τις πληροφορίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Δεν έχουμε ακόμα ε, πλήρη ανάπτυξη συστήματος, αλλά έχει κάπως ξεκινήσει. είναι ένα κράτος μέλος ελέγχει ένα προϊόν, ενώ, ενώ ένα άλλο κράτος μέλος ε, δεν το ελέγχει, τότε έχουμε κάποια τριβή με συνέπεια κενό ασφαλείας. Γιατί σε περίπτωση πραγματικής απειλής ασφάλειας μπορεί να περάσει. Αφετέρου δεν έχουμε και πρόβλημα ως προς τον ανταγωνισμό γιατί στο μεν κράτος περνάει χωρίς άδεια ενώ στο άλλο μπορεί να περάσει μόνο με άδεια. Και το ίδιο θα συνεχίσω με τις ενδοκοινωτικές μεταφορές, ενδοομιλιακές μεταφορές, αλλά αυτό το κάλυψα. Εφαρμογή και υλοποίηση αποτελεσματική. Σημαντικό θέμα. Είμαι πεπισμένος εδώ ότι ο μηχανισμός και η βελτίωση της, ε, του διοικητικού πλέγματος γύρω από την ε, ρύθμιση είναι εξίσου σημαντική με τη ρύθμιση. Έχουμε δηλαδή ένα σύστημα οικονομικό διπλής χρήσεως που λειτουργεί, ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο, το οποίο μας στηρίζει στην ανταλλαγή πληροφοριών και έχουμε μάλιστα προχωρήσει αρκετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύστημα αυτό. Ε, η βασική ιδέα είναι να διατίθεται σε όλα τα κράτη-μέλη ε, να διατίθενται ε, οι ηλεκτρονικές άδειες που έχουν ήδη στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες των κρατών μελών, των λοιπόν κρατών μελών, αλλά ίσως θα πρέπει να διευκρινίσουμε περισσότερο αυτή την ιδέα σιγά σιγά. Κάτι άλλο, ε, γιατί οι έλεγχοι των διπλών χρήσεων, των προϊόντων διπλής χρήσεως αφορούν τους πάντες και τις υπηρεσίες αντιοδότησης αλλά και τα τελωνία και μάλιστα πολλές φορές ένας υπάλληλο τελωνίου ε, μπορεί να μην έχει επαρκή κατάρτιση μόνο και μόνο γιατί η χώρα του δεν παράγει το συγκεκριμένο προϊόν διπλής χρήσης. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η κατάρτιση, χρειάζεται και η επαφή με υπαλλήλου ε, με στελέχη τρίτων χωρών που πρέπει να μας ενημερώσουν για τη διπλή χρήση. Έχει τεράστια σημασία για μας. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αναλάβουμε πιο διαρθρωμένη δράση και εσωτερικά. Και ένα τελευταίο σημείο, όπως είπα, η έλεγχη των εξεγωγών προϊόντων διπλής χρήσης σημαίνει εμπλοκή και συμμετοχή των πάντων. Δεν μπορούμε, να ξεκινήσουμε, δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε αποτελεσματικότητα χωρίς τη σύμπραξη και του κλάδου παραγωγής, όπου θα θέλαμε την συμμόρφωση σε προδιαγραφές ως κριτήριο απαραίτητο για την ε, εξασφάλιση φερρυπίν ε, μιας συλλήβδην άδειας. Και αντίστοιχα θέλουμε να διασυνδέσουμε αυτή τη ε, συμμόρφωση με άλλα συστήματα όπως το σύστημα των τελωνίων ε, για την ε, δυνατότητα διοδότηση των εξαγωγέων κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μελετάμε με ομάδες εργασίας στο Συμβούλιο και εν Διαφάνεια, έχουμε την ετήσια έκθεση διαφάνειας. Τη διαβιβάσαμε μάλιστα πριν από μερικά λεπτά μόλις. Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ελέγχους προϊόντων διπλής χρήσεως ε, με στόχο να ενημερώσουμε τους χρήστες και το κοινό. Ξέρουμε ότι δεν θα μείνουν ποτέ αυτά τα πράγματα κρυφά, αλλά θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί εάν μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και χάρη στους κατασκευαστές και εξαγωγείς. Προσπάθησα να ολοκληρώσω το χέτερο δυνατό, είναι όμως τόσο ευρύ το θέμα και ως συνήθως μακρηγόρησα. Ζητώ συγγνώμη, εκ των προτέρων λέει ο μιλητής, επειδή ξεπέρασα ήδη το χρόνο μου. Πολύ ευχαριστώ να ακούσω οποιασδήποτε ερωτήσει ή παρατηρήσει και επίση ευχαριστώ ιδιαίτερα στι δύο επιτροπέ που συνοργάνωσαν τη συνεδρίαση για την ευκαιρία να συλλέξουμε εμπειρίε και προτάσει. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκαρτσότη για την πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά του. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Στιούαρτ από το King's College. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίσης ευχαριστώ την Επιτροπή και την Υποεπιτροπή για την πρόσκληση να βρεθώ σήμερα εδώ μαζί σας. Τώρα, όσον αφορά στο υπόβαθρό μου και την καριέρα μου που έχει σχέση εδώ με τις παρατηρήσεις μου, να πω ότι ήμουν υπεύθυνος για τις για την εφαρμογή μίας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν περάσω πριν από τέσσερα χρόνια στον τομέα της πάταξης ε, της μετάδοσης του εμπορίου. Να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος της λεπτομέρειας, μ' αρέσει η επικοινωνία και οι αρχές ε, και προσπαθώ να καταλάβω πέρα από τις αρχές τις λεπτομέρειες για τις οποίες μιλάμε. Ο τρόπος που έχω διαρθρώσει τις παρατηρήσεις μου ε, έχει να κάνει με τέσσερες ε, τομείς προτεραιότητας ε, και με βάση αυτούς θα κάνουμε την παρουσίαση. Ας πάμε στην πρώτη διαφάνεια. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας σημαντικός παραγωγός προϊόντων διπλής χρήσης. Να το ποσοτικοποιήσω κάπως. Υπάρχει σημαντικό θέμα για τη συλλογή δεδομένων σε αυτό το τομέα και δυστυχώς δεν έχουμε μια καλή εικόνα για το τι παράγεται ούτε στην Ευρώπη ούτε παγκοσμίω. Γενικά όμως ε, μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παραγωγούς ευαίσθητης τεχνολογίας σε επίπεδο διάδοσης ε, ε, όπλων. Και πάντοτε ε, ε, στην ιστορία ήταν στόχος των ανθρώπων ε, που ασχολούνταν με αυτό το θέμα. Το 1978 είχαμε το πρώτο παράδειγμα ε, διπλής χρήσης προϊόντων με ένα πρόγραμμα ε, που υπήρχε τότε και έκτοτε έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος. Ε, ο, ο χρόνος βέβαια δεν βοήθησε στο να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα πλήρως. του λεχθέντος η ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι κανονισμοί έχουν γίνει πολύ καλοί. Ειδικότερα όσον αφορά στην ενημέρωση των καταλόγων και πολλά ζητήματα έχουν επιλυθεί οπότε σίγουρα δεν χρειάζεται να αρχίσουμε εκ του μηδενός υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα να ε, χτίσουμε πάνω στο πλαίσιο που ήδη υφίσταται έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η δουλειά μας. Και όταν λέω πιο αποτελεσματική μπορούμε να είμαστε πιο στοχευμένοι και ε, αυτό ε, σημαίνει ότι θα είμαστε και πιο χαλαροί σε κάποιους τομείς. Ένα βασικό στιγμίο εδώ είναι ότι η εφαρμογή ποικίλει ανάλογα με το κράτος. Όντως φαίνεται πως αυτό είναι το πιο ε, επίγον θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών. Και πραγματικά ε, εκτιμώ τη δουλειά που έχει γίνει εκτός Ευρώπης για ε, τους ελέγχους σχετικά με τις εξαγωγές και τις δυνατότητες και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο σε αυτό το τομέα εσωτερικά. Ένα άλλο βασικό σημείο εδώ είναι ότι πολλές χώρες εκτός Ευρώπης κοιτάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τη βάση για τους δικούς τους ελέγχους εξαγωγών, είτε χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες λίστες, είτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των κανονισμών. Και θα πήγαινα ακόμα πιο μακριά και θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι η ηγετική σημασία γιατί Όλοι κοιτάνε αυτή την νομοθεσία, οπότε ε, πέρα από ευρωπαϊκή νομοθεσία τελικά έχει καταλήξει να γίνει ένα παγκόσμιο στάνταρ, ένα παγκόσμιο πρότυπο. Τώρα, δεν θα μπω ε, σε λεπτομέρειες σχετικά με τους κανονισμούς και το θέμα του ελέγχου των εξαγωγών. Να πω όμως ότι θα πρέπει κανείς να δει τι κάνει κάθε χώρα σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων. Και πρέπει πραγματικά να πούμε ότι σε κάποια μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η τάση να εξετάζονται πρώτα οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, το καταλαβαίνω, αλλά όταν κοιτούμε τις λεπτομέρειες η εικόνα είναι διαφορετική. Στη ΣΥΠΑ οι μεταρρυθμίσεις έχουν να κάνουν με το δικό τους ιστορικό πλαίσιο και συγκεκριμένα με το πώς ελέγχουν τα στρατιωτικά αγαθά και πώς δίνουν διάφορες άδειες ε, στους οργανισμούς τους. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχουν ε, τροπολογίες οι οποίες κατατίθενται στις ΕΠΑ για αυτό το λόγο και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία παραμένει πολύ ανταγωνιστική σε αυτό το πλαίσιο. Τούτου λεχθέντως να πω ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πολύ συχνά ακούω να λέγεται ότι είναι πολύ καλές ε, ε, μεν, αλλά ανταγωνίζονται πολύ τη ΣΥΠΑ ως προς την ενιαία άδεια που έχουν για τις επιχειρήσεις. Όταν μίλησα με Αμερικανούς για το σύστημά μας ε, μου είπαν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε ένα εξαιρετικό σύστημα και μπορείτε να κάνετε τόσα ε, ωραία πράγματα με αυτόν τον κανονισμό που έχετε που εμείς δεν μπορούμε. <laughs> Τελικά ε, φαίνεται ότι το βότι του γείτονα είναι πάντα πιο παραγωγικό. Έτσι λοιπόν πάμε στην επόμενη διαφάνεια και να πω ότι... Υπάρχει όντως μεγάλη δυσκολία να ποσοτικοποιήσουμε τα αγαθά που ελέγχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα έγινε μια μελέτη για αυτό το θέμα και καταλήξαμε με ένα νούμερο ε, που είναι γύρω στα 26 με 36 ε, δις. Ε, πραγματικά δεν είναι εύκολο να δώσουμε συγκεκριμένη απάντηση. Αυτό που κάνουμε λοιπόν στο Kings είναι ε, να κάνουμε μια έρευνα η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα ε, θέματα. Στα αριστερά βλέπετε τους παραγωγούς ε, τεχνολογίας υψηλής τεχνολογίας και βλέπετε πόσο μεγάλη συγκέντρωση υπάρχει στην Ευρώπη. Όταν όμως κοιτάμε τη δεξιά εικόνα βλέπουμε τι γίνεται με τις μεταφορές, τη διαμετακόμιση. Ένα γράφημα λοιπόν το οποίο δείχνει ότι κυρίως η Κίνα είναι ε, ο ηγέτης σε αυτό το τομέα. Βέβαια, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλό θα ήταν να συνεργαστούμε ώστε να έχουμε ένα χρωματικό σύστημα το οποίο θα είναι τόσο λαμπερό όσο και στις άλλες χώρες. Ε, θα δούμε λοιπόν αν αυτό μπορεί να γίνει στο μέλλον. Πάμε τώρα να πούμε για τις τέσσερις αρχές. Όπως είπα, Υποστηρίζω τις αρχές της ανακοίνωσης, εγώ όμως ασχολούμαι με τις λεπτομέρειες, τις παίρνω και τις εξετάζω. Όσον αφορά στην ανθρώπινη ασφάλεια, είναι ένας όρος ε, με τον οποίο όλοι συμφωνούμε, όμως αυτό τι σημαίνει στην πράξη, αναρωτιέμαι. Να ελέγχουμε επιπλέον τεχνολογίες ε, σημαίνει να προσπαθούμε να μην ε, εξάγονται οι τεχνολογίες σε κάποιους συγκεκριμένους τόπους και αυτό πώς διαφέρει από τις κυρώσεις. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο των εξαγωγών πραγματικά ε, πολλές φορές με δυσκολεύει. Δεν μπορώ να το ε, διαχωρίσω από τις κυρώσεις. Πρέπει λίγο να δούμε ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε διαθέσιμα για να τα συνδυάσουμε. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε γενικότερες στρατηγικές που θα καλύπτουν τα πάντα σε αυτό το τομέα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται ε, από άποψη στρατηγικών στόχων, πέρα από τους ελέγχους, να δούμε ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε και να τα χρησιμοποιούμε. Τώρα, για την έξυπνη ασφάλεια. Επειδή έχω αυτή την ανησυχία για τις διαφορές στην εφαρμογή στην κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προκλήσεις ε, που αυτό ενέχει για τις μικρότερες χώρες που δεν έχουν ανθρώπινο δυναμικό και άλλων μορφών πόρους, να πω ότι αυτό επηρεάζει και το δικαίωμα ε, στην πρόσβαση στην εμπειρογνωμοσύνη και ούτω καθεξής. Οπότε, αυτό έχει να κάνει και με το καθεστώς ελέγχου των ε, ε, εξαγωγών. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα και θα σας πω στα συμπεράσματά μου κάποια στοιχεία, κάποιες σκέψεις ε, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια. Γιατί εδώ έχουμε ε, έναν τομέα με πολύ μεγάλη ρύθμιση. Έχω στο Kings ασχοληθεί πολύ με τον έλεγχο των εξαγωγών και έχω μάλιστα εκδώσει και έναν οδηγό. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι, ποιοι είναι οι ορισμοί για τη βασική επιστημονική έρευνα στο δημόσιο χώρο κτλ. Υπάρχουν ε, πρακτικά ζητήματα σε αυτούς τους ελέγχους λοιπόν. Επίσης ενοιολογικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, το τι κάνουμε σε σχέση με τον έλεγχο των υλικών. Ας πούμε με τη τριδιασδιάστατη εκτύπωση πώς θα καταλάβουμε και πώς θα πιάσουμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, ε, πώς ε, θα ε, γίνεται μεταφορά των δυνατοτήτων στις άειλες τεχνολογίες, κάτι που δεν υπάρχει σε κάποιο διάγραμμα και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τεράστια παρουσίαση για τις διάφορες μορφές γνώσης σε αυτόν τον τομέα. Προσπαθώ λοιπόν να σκεφτώ πιο ενοιολογικά το ζήτημα του ελέγχου των υλικών. Διότι ε, αυτό όντως φαίνεται ότι πάει πέρα από τον κανονισμό για τον έλεγχο των εξαγωγών. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Το είπα και αυτό πριν, δεν θα επεκταθώ, αλλά η εφαρμογή ποικίλει από κράτος σε κράτος. Μιλήσαμε για τις προκλήσεις σχετικά με την εφαρμογή σε επίπεδο πρακτικό στις άδειες. Κάποια ε, κράτη προσφέρουν ανοιχτές ε, άδειες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι. Ειδικά αυτός ο τομέας πραγματικά έχει ε, μεγάλο δυναμικό για να υπάρξουν στρεβλώσεις μεταξύ των χωρών. Επόμενη διαφάνεια. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν σε σχέση με τις ανοιχτές άδειε για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε λίγο από αυτές τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια. Έχω συγκεκριμένες ιδέες γι' αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν δυνατότητες, νομίζω σε τρία διαφορετικά πλαίσια, για να σκεφτούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις ανοιχτές άδειε πιο ευέλικτα, να υπάρχει μία προσέγγιση βάση της τιμής. Δεν εννοώ ε, ας πούμε ε, εμπορεύματα χαμηλής αξίας, θα πρέπει απλώς να δούμε τι εμπορεύματα είναι αυτά που ελέγχουμε και βάσει αυτών να ρυθμίζουμε ε, την προσέγγισή μας. Τώρα, ο χάρτης αυτή την εικόνα δείχνει ε, μια ανάλυση των δεδομένων των αδειών στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από μερικά χρόνια. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες 0, 1, 2, 3, 4 και ούτω καθεξής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε κατηγορία 5 για αυτές τις άδειες, είναι το πράσινο χρώμα και είναι αυτό που προεξέχει σε επίπεδο αξίας, ε, αυτό που ε, είναι πιο δημοφιλές. Μπορούσαμε να μιλήσουμε ώρες γι' αυτό. Πάμε τώρα λοιπόν στην προσέγγιση βαστών κινδύνων. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ποτέ θα φτάσουμε στη θέση ώστε κάθε κράτος μέλος να έχει τα ίδια συμπεράσματα για κάθε άδεια. Είναι δύσκολο. Όμως υπάρχουν δυνατότητες σύγκλησης, να υπάρχουν πιο πολλά κοινά στοιχεία σχετικά με τις αποφάσεις για τις άδειες. Και όσον αφορά αυτό το θέμα, ε, δηλαδή την εκτίμηση κινδύνου και τα κριτήρια, υπάρχει κανονισμός ο οποίος αφήνεται στα κράτη-μέλη την ε, διακριτική ευκαιρία να βγάλουν δικά τους κριτήρια συγκεκριμένα ε, ε, ε, επίσης να χρησιμοποιήσουν κριτήρια που προτείνονται από τον κανονισμό, ε, έτσι ώστε να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος κατάλογος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των αδειών. Όσον αφορά στην ασφάλεια των ανθρώπων, νομίζω ότι τα κριτήρια αυτά ε, θα ήταν ένας τρόπος να ενσωματώσουμε αυτή την αρχή στις αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη. Και υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά στο να έχουμε κοινούς ε, κανόνες. Θα το πω λίγο καλύτερα αργότερα. Τώρα, να πω για τις μεταφορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα θέματα που είναι πολύ ε, δημοφιλή. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, ε, άδειε που απαιτούνται ακόμα και για τη μεταφορά προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες να μειωθούν οι απαιτήσει. Βέβαια, είναι σημαντικές οι απαιτήσει γιατί ε, πρέπει κανείς να γνωρίζει ότι τα προϊόντα θα μπορούν να εγκρίνονται και από εξωτερικούς φορείς. Ε, συνεπώς, ε, καλό είναι να υπάρχει μια δυνατότητα υποστήριξης. Το μόνο θέμα εδώ, στο οποίο θα δίσταζα, θα ήταν το να αλλάξουμε τα συστήματα ώστε να προσαρμοστούμε σε μια σειρά από διαφορετικές μικρές επιχειρήσεις που θα έχουν διαφορετική φωνή και ε, τοποθετήσεις. Θα χρειαστεί μια σειρά από γενικού τύπου νομοθεσίες ώστε να έχουμε τις επενδύσεις στο τομέα αυτών. Στην επόμενη διαφάνεια, αν κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνοχή και την παραγωγή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό αυτό της ανταλλαγής πληροφορίας. Και εδώ δεν εννοώ μόνο κοινοποιήσεις που θεωρείται ότι είναι η στάνταρ μορφή επικοινωνία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας και ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Τα συστήματα ελέγχου των εξαγωγών έχουν τόσο ή άλλως πολύ αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να ε, ελέγχουν και να επαληθεύουν τις ανταλλαγές, απλώς, τις συναλλαγές. Απλώς δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην Ευρώπη ίσως μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα. Και πρέπει να εναποτεθεί αυτή η λύση στον έλεγχο των εξαγωγών. Στην επόμενη διαφάνεια επανέρχομαι στις αρχικές μου παρατηρήσεις ότι το πεδίο ανάπτυξης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ε, θα είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε εταίρους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμορφωθούν με τις δικές μας προτάσεις, αν εμείς με στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε καταλήξει σε ένα καλό επίπεδο συνεργασίας. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ε, καλό πρόγραμμα εσωτερικό για την αδειοδότηση και την κοινοποίηση γνώσης και πληροφορίας. Και θα πάω στο επόμενο στην επόμενη διαφάνεια. Ζητήματα της ε, άδειας είναι πολύ σημαντικά. Όταν φτάσουμε στο σημείο εξόδου στα σύνορα, αντί να προσπαθούμε σαν αντίληψη να παρεμποδίσουμε την εξαγωγή του προϊόντος στο, από τα σύνορα, ε, πρέπει να κοιτάξουμε μία, μία σειρά ε, παραγωγής, μια αλυσίδα παραγωγής. Και γι' αυτό θα ήθελα εδώ να καλωσορίσω και την ε, κοινοποίηση για την συμπερίληψη στις προσπάθειες της στρατηγικής σημασίας βιομηχανίας. Αυτή η συμπερίληψη δεν πρέπει απαραίτητα να προκύψει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχει να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να δουν ε, με μια ολιστική προσέγγιση τους κινδύνους τους οποίους εκτίθενται. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερος το την πρόταση κατευθυντηρίων γραμμών που είδαμε πρόσφατα, ε, που θα μπορούσε ε, ε, προερχόμενη από, την, από τους προμηθευτές, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορίσαμε λοιπόν τα, τους τομείς προτεραιότητας. Εγώ νομίζω ότι είναι καλή η ευρωπαϊκή νομοθεσία χωρί βελτίωσης όμως με ένα σύστημα εσωτερικής προσέγγισης μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να κάνουμε πολλά επίσης προς την κοινή αξιολόγηση κινδύνου, κοινά κριτήρια και ούτω καθεξής. Και βεβαίως οι ατόμων όπως και η έλεγχοι των εξαγωγών θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, αλλά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους ελέγχους εξαγωγών για το στόχο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα η δόκτωρ Σιμπίλ Πάουερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μου δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρω και εγώ σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική συζήτηση και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια προσωπική παρατήρηση. Ε, ήμουν πολύ καιρό εδώ όταν έγραφα την διδακτορική μου διατριβή για τους ευρωπαϊκούς ελέγχους ε, ε, των εξαγωγών και τη δυνατότητα ελέγχου από πλευράς ε, κοινοβουλίων. Βλέπουμε ότι τα θέματα αυτά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και στο θεματολόγιο των ε, κοινοβουλίων και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που το, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται τόσο επί του ζητήματος. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που έχουμε να καλύψουμε εδώ σε αυτό το εργαστήριο με πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, γι' αυτό θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε κάποια από τα ουσιαστικά σημεία. Ήδη ε, είχαμε μία εικόνα των ε, δυνατοτήτων αναθεώρησης από τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο συνάδελφος ο Ιαν Στιούαρτ ήδη επεσήμενε κάποια από τα βασικά στοιχεία των ελέγχων των εξαγωγών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες δυνατότητες αναθεώρησης. Θα έχετε δει ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φυσικά εσείς μπορείτε κάλλιστα να θίξετε και άλλα θέματα στη διάρκεια της ε, συζήτησης που θα γίνει μετά τις παρουσιάσεις. Θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να δούμε λίγο τον τίτλο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος τίτλος λέει ότι η αναθεώρηση της πολιτικής γίνεται προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια σε έναν ε, ολοένα ε, εναλλασσόμενο κόσμο. Και επομένως εδώ τίθεται θέμα ελέγχου εξαγωγών Τι προσπαθούν να κάνουν οι έλεγχοι των εξαγωγών. Προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει ασφάλεια και ανθρώπινη ασφάλεια αλλά και ασφάλεια εν γέννη και να έχουμε ισορροπία μεταξύ οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων. Και το βλέπουμε αυτό διότι υπάρχουν δύο διαφορετικές επιτροπές ε, και υποεπιτροπές οι οποίες ε, φιλοξενούν το συγκεκριμένο εργαστήριο υπάρχει το θέμα που έθιξαν και οι συνάδελφοι, των άιλων μεταφορών τεχνολογίας και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να προσθέσουμε και μια τρίτη διάσταση. Να εξισορροπήσουμε τους ελέγχους των εξαγωγών με την ε, ακαδημαϊκή ελευθερία. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία είναι εξελίξη αυτή τη στιγμή. Ε, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να επιβάλλουμε περιορισμούς ε, κατά την ακαδημαϊκή ανταλλαγή πληροφοριών όταν αυτά σχετίζονται με ε, ευαίσθητες ε, τεχνολογίες από πλευράς ασφαλείας ε, εν γέννη. Το πρώτο θέμα λοιπόν το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι κάτι το οποίο τονίζεται ιδιαίτερα στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις άειλες μεταφορές τεχνολογίας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με δύο τρόπους, είτε μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας, αλλά και μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης. Επομένως, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες οι οποίες αναρτώνται σε κάποιον ε, σερβερ. Και εάν κάποιος αναρτήσει πληροφορίες σε ένα σερβερ, αυτό σημαίνει ότι διατίθεται και μπορεί κάποιος να τις χρησιμοποιήσει, να τις κατεβάσει σε μια άλλη χώρα. Επομένως, εσείς συμμετέχετε σε μια εξαγωγή. Η ανταλλαγή πληροφοριών, λοιπόν, ε, όταν αναφερόμαστε σε εξαγωγή και έλεγχο των εξαγωγών ε, έχει αλλάξει πάρα πολύ και έχουμε μεταφερθεί πολύ από την παραδοσιακή εξαγωγή ε, αγαθών. Δεν υπάρχει τελωνιακός υπάλληλο ο οποίος μπορεί να ελέγξει την εξαγωγή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την ανάρτηση πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή των ελέγχων εξαγωγών έχει αλλάξει άρδιν από την ε, εξέλιξη της τεχνολογίας. Έχουμε τη συντομογραφία ITT για την άλλη μεταφορά τεχνολογίας και αυτά τα ITTs είναι πολύ σημαντικά για τις ανταλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Έχουμε ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων, κυρίως πολυεθνικών επιχειρήσεων, ανθρώπους που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο με λάπτοπ που έχουν τεχνολογία ε, εντό και το θέμα είναι πότε μπορεί κάποιο να ζητήσει άδεια, όταν πάει σε ένα συνέδριο, όταν φεύγει από το συνέδριο, όταν φτάνει στην επιχείρηση και το καθεξής. Και επίσης το ITT είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ακαδημαϊκή έρευνα. Δεν μπορεί να γίνει ακαδημαϊκή έρευνα έρευνα χωρίς ανταλλαγή γνώσεων και χωρίς δημοσιεύσεις. Και υπάρχει και το ερώτημα σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνονται έλεγχοι για τις δημοσιεύσεις και αυτό σχετίζεται με το ITT όταν αφορά μεταφορά τεχνολογίας. Από τις διαβουλεύσεις τις οποίες συμμετείχαμε για το σχέδιο συλλογής δεδομένων που είχαμε, διαπιστώσαμε ήδη ότι υπάρχει σαφώς ανάγκη και έτοιμα για διευκρινήσεις αλλά και πρακτικές ε, κατευθύνσεις στον τομέα του ITT. Τώρα, να περάσουμε σε ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο τόνισαν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, το θέμα της δημιουργίας δυνατοτήτων. Δημιουργία δυνατοτήτων και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς. Αυτό το οποίο επεσήμανε ο Ιαν Στιούαρτ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να το τονίσω και πάλι. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας προπολογισμό ε, για ε, εσωτερικές ε, δημιουργίες δυνατοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό μας έχει οδηγήσει σε μια παράλογη μάλλον κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιες δυνατότητες οι οποίες χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι είναι μια σειρά από σεμινάρια και δραστηριότητες που διεξάγει στην Ευρώπη το πρόγραμμα ελέγχου των εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως με χώρες οι οποίες προσφάτως εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτάχρονα δαπανώνται ουσιαστικά ποσά ε, για την ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ελέγχους σε τρίτες χώρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχει προσδώσει μεγάλη ουσία και στην ασφάλεια αλλά και στην ενίσχυση της παγκόσμιας σύγκλησης και να έχουμε ισότιμους αίρους ανταγωνισμού. Αυτό που προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά σημαντικό σε θέματα δημιουργίας δυνατοτήτων και εσωτερικής κατάρτισης και δεν αφορά μόνο τη διαδικασία διοδότησης αλλά περιλαμβάνει και το όλο φάσμα της εφαρμογής όλων αυτών των λειτουργιών. Και επίσης πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι ε, και η εσωτερική και η εξωτερική προσέγγιση ενισχύουν η μία την άλλη. Εάν λοιπόν ενισχύσουμε την εσωτερική προσέγγιση, αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού για τα προϊόντα διπλής χρήσης, κάτι το οποίο ανέφερα και προηλαλήσαντες, αλλά πρέπει να πω ότι και από τη δική μου τη σκοπιά η διαφορετική εφαρμογή δεν είναι κάτι απαραίτητο αρνητικό, διότι χρειαζόμαστε διαφορετικά συστήματα σε κάθε χώρα. Τα πάντα βέβαια θα πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι μια σημαντική διάκριση η οποία πρέπει να γίνει. Μία τρίτη παρατήρηση, η οποία αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η ενισχυμένη στρατηγική και επιχειρησιακή συνεργασία με τις οργανισμούς επιβολής ε, και εφαρμογής. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών των οργανισμών και εδώ υπάρχει μια κάπως παράλογη κατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει ένα ε, διαρθρωμένο σημείο επαφής για τους οργανισμούς αδειοδότησης και για πολλά από τα Υπουργεία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν υπάρχει ένα θεσμικό βήμα αυτή τη στιγμή όπου αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα εφαρμογής θα μπορούν να συναντώνται και να συζητούν τα της εφαρμογής της Βρυξέλλες σε τακτική βάση. Υπήρχε μια συνάντηση κάποια στιγμή, αλλά δεν συνεχίστηκαν οι επαφές σε τακτική βάση και αυτό σημαίνει ότι αν οι αρχές εφαρμογής ασχολούνται με τον έλεγχο, την πρόληψη, τον εντοπισμό, την έρευνα, τη δίωξη και θέλουν να ανταλλάξουν πληροφορίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ συχνά θα πρέπει να γίνεται σε συναντήσεις ε, διεθνείς, σε εκδηλώσεις στη Σιγκαπούρη ή στην Ουκρανία ή θα πρέπει να γίνονται σε συνεδριάσεις που χρηματοδοτούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και ένα άλλο θέμα εδώ. Είναι μία πρόταση ότι δεν μπορεί η Επιτροπή να ορίσει προτεραιότητες πολιτικής, εποκύκλους επιτροπη να ορισει προτεραιοτητες πολιτικης ποκυκλους πολιτικης όπου εγώ δίνω την εξή ε, ερμηνεία, ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει έλεγχος εξαγωγών κατά προτεραιότητα για τους διάφορους τομείς θεσμικής αρμοδιότητας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα από τα πιο ε, ακανθόδη ζητήματα, δηλαδή ότι μερικές φορές μείνει ανάμεσα σε δύο καρέκλες ο έλεγχος εξαγωγών ε, δι, του, ε, δι της Δεν είναι κανείς αποκλειστικά αρμόδιος για να ελέγξει τις εξαγωγές. Και εδώ πολύ συχνά ρυθμίζουν την κατάσταση ή τα Υπουργεία των Εξωτερικών ή τα Τελωνία. Η κατάσταση όμως στην πραγματικότητα στην Ευρώπη σήμερα αλλά και στα περισσότερα μέρη του κόσμου είναι ότι τα τελωνία προτεραιότητα έχουν τις εισαγωγές και την περισυλλογή εσόδων. Όχι ε, ασφάλεια και όχι έλεγχο εξαγωγών. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουν προτεραιότητες για μια πιο ουσιαστική Εκεί πρέπει να γίνει η αλλαγή λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Και νομίζω επίσης ότι αυτό που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε αν προκειμένου είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας με τους φορείς του έχει επίσης αλλάξει η μορφή σε σχέση με την πολιτική ελέγχου των εξαγωγών. Υπήρχε ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγωγές, άρα πρέπει να στραφούμε προς τις εξαγωγές πάντα, αλλά με τους ελέγχους στη διαμεσολάβηση, την δια ε, διέλευση την δια, ε, ε, ή την μεταφόρτωση και την διαβίβαση γνώσεως πρέπει να στραφούμε και προς τον χώρο των ερευνητών, ακαδημαϊκών, μεταφορέων και το καθεξής και γι' αυτό Ιδιαίτερη έμφαση ε, πρέπει να δοθεί στην τρισδιάστατη εκτύπωση που προβάλλεται ε, και μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επίδραση και στον χώρο των μεταφορών. Οι μεταφορές, από ό,τι λέγεται σιγά σιγά, στο μέλλον θα γίνονται με τρισδιάστατη εκτύπωση. Ένα άλλο θέμα βέβαια στο οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε με προσοχή είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινα η ασφάλεια, των ανθρώπων, γιατί εδώ έχουμε μια ουσιαστική αλλαγή. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με προϊόντα διτά, έτσι, ε, πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης. Αλλά πρέπει να προσθεθεί και μια τρίτη διάσταση. Η πιθανολόγηση χρήσης τους σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ε, σε αμφισβήτηση της ασφάλειας των ανθρώπων. Άλλο σημείο σημαντικό είναι η βασική έννοια της εξαγωγής και του εξαγωγέα. Όπως έχει τώρα ο κανονισμός, ιδιαίτερη έμφαση και εστίαση δίνεται στον εξαγωγέα. Είχε αλλάξει όμως η πραγματικότητα. Ιδιαίτερη σημασία λοιπόν έχει ως φορέας αυτός ο οποίος εμπλέκεται στην διαμετακόμιση ή διέλευση ενός προϊόντος. Δεν ξέρουμε ποιο είναι, αλλά έχει σημασία το ότι υπάρχει αυτή η διέλευση και πρέπει αυτό το στοιχείο να αντιμετωπιστεί νομικά. Αυτά είναι νομίζω από την επισκόπηση τη δική μου και για να συνοψίσω κλείνοντας κάποια από τα κύρια σημεία, προχωρώντας αυτό που θα πρέπει να προσαρμοστεί θα είναι καταρχάς η, μετάβαση από η μετάβαση από την παραδοσιακή προσέγγιση μεταξύ και διάκριση μεταξύ, μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης στην ε, διάσταση προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ασφάλειας του ανθρώπου. Μετά, μετάβαση από τη διάκριση εξαγωγών, εισαγωγών, ε, εξαγωγών, εξαγωγέα καλύτερα στις λοιπές διαστάσεις, διαμετακόμιση, διέλευση, μεταφορά κτλ. Ε, υλικά άειλα αγαθά που μας ε, επιβάλλει άλλωστε η τεχνολογική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει επίσης να δοθεί στη διατήρηση των εξωτερικών συνεπειών για τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις δηλαδή σε αυτές αλλαγές, όπως άλλωστε είπε και ο προλαλής σας, και πρέπει ιδιαίτερα το κοινοβούλιο σας όταν συζητεί θέματα της ε, βελτίωσης της διαδικασίας για την αναθεώρηση του ελέγχου, του καταλόγου ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνειδητοποιεί και να παρακολουθεί και συζητήσεις που γίνονται στον υπόλοιπο κόσμο, στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Μαλαισία και με τον κυβερνήτη της Σιγκαπούρης έτυχε να συνομιλήσω που μου λέγανε πότε θα γίνει αυτή ο κατάλογος των ε, Ευρωπαίων επιτέλους να είμαστε έτοιμοι και εμείς γιατί εμείς παρακολουθούμε αυτά που αποφασίζουν οι Ευρωπαίοι. Όταν έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια λειτουργία προτύπου για άλλε χώρε του κόσμου, στα διάφορα στοιχεία, οτιδήποτε αποφασίστε στι Βρυξέλλε, ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλε συνέπειε για τα συστήματα άλλων κρατών και αυτό σημαίνει πολύ σημαντική ευθύνη ταυτόχρονα για μένα. Τέλος, η σημασία την οποία υπενήχθην ε, στην αρχή, αλλά έχει νομίζω λόγο να την επαναλάβω, ε, το, το, ότι είναι εύκολο βέβαια να ορίζουμε προτεραιότητες, στρατηγικές πολιτικές προ, ε, προτεραιότητες, να διαθέτουμε πόρους για την υλοποίηση όμως και η πραγματική υλοποίηση είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε μεγάλες προκλήσεις ως προς την υλοποίηση και την τήρηση των προδιαγραφών του ευρωπαϊκού δικαίου σήμερα. Αυτό σημαίνει διάθεση επαρκών πόρων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αρκετό χρήμα αυτή τη στιγμή για προσωπικό, όπως απαιτείται, κυρίως ε, στο δυναμικό ε, επίβλεψη της στήριξης του νόμου, τελωνιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες των Υπουργείων Ιστορικών κτλ. Και βέβαια υπάρχει ανάγκη για την κινητοποίηση πόρων, για την εσωτερική συνεννόηση και διευθέτηση, ε, όπως απαιτείται. Ευχαριστώ και έτσι κλείνω και δίνω το λόγο πάλι στην Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για τα πρακτικά της σημερινής συζήτησης. Προτείνω, λοιπόν να λάβει το λόγο ο κύριος Βίνκλερ πρώτα για να κάνει κάποια σχόλια για τις παρουσιάσεις και δεχομένως να διατυπώσει ερωτήσεις ε, από την προοπτική της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου έτσι ώστε και οι συνάδελφοι που είναι παρόντες στην αίθουσα να διατυπώσουν με τη σειρά τους τις ερωτήσεις τους. Και θα ήθελα και εγώ να λάβω το λόγο για να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις, να ολοκληρωθεί έτσι ο πρώτος γύρος και μετά θα παρακαλέσω τον κύριο Βίνκλερ να αναλάβει το δεύτερο γύρο εφόσον μας το επιτρέψει ο χρόνος βέβαια, θα ακουστούν και ερωτήσεις από το κοινό. Σε ένα δεύτερο όμως γύρω ερωτήσεων. Κύριε Βίγκλερ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μακρηγορήσω. Θα διατυπώσω όμως κάποιες παρατηρήσεις για να δώσω στη συνέχεια το λόγο στους συναδέλφους της ε, στον συνάδελφο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, τον κύριο Κέλαμ. Πρώτη μου παρατήρηση λοιπόν, ότι έχουμε να κάνουμε με θέματα ε, διεπιστημονικά, διατομεακά και που αφορούν βεβαίως και τις εργασίες της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Τη στιγμή που μιλάμε έχουμε συναφή ζητήματα εκρεμή ε, επί παραδείγματι της, ε, την διακίνηση ορισμένων ε, προϊόντων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ε, προσβλητική, υποτιμητική ε, μεταχείριση, προσβολή της προσωπικότητας, βασανιστήρια, ακόμη και θανατικές ποινές. Συναφή λοιπόν τα ζητήματα. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν μπορούμε να δεχθούμε ότι υπάρχει ανάγκη για μια πιο ενοποιημένη, ολοκληρωμένη προσέγγιση πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεχθούμε, γιατί νομίζω ότι είναι και προφανέ, ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων περιοχών των ελέγχων των εισαγωγών, των εξαγωγών. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε περισσότερη συνοχή, εναρμόνιση και ολοκλήρωση, μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωση μεταξύ των διαφόρων αυτών τομέων, δηλαδή διπλή χρήση υλικά για τη βασανιστήρια, τρομοκρατία και το καθεξής. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την, ε, την παρουσίαση του κυρίου Κατζότη και βλέπω ότι μιλάτε σαν τίτλο για τις εξελίξεις σε έναν μεταλλασσόμενο κόσμο. Ίσως λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε, γιατί βλέπω ότι αντίστοιχη προσέγγιση, ότι έχουμε να κάνουμε μια νέα πραγματικότητα, είχαν και οι άλλοι ομιλητέ. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι στο τίτλο σας ήταν προσφορότερο να ονομαστεί ε, υλικά διπλής χρήσης σε έναν ταχύτατα μεταλλασσόμενο κόσμο. Δεν έχουμε πια τόσο πολύ χρόνο για προσαρμογή και εξυγχρονισμό της νομοθεσίας μας, η επικαιροποίηση. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι το εξής, μια και όλοι οι, ομιλητές, οι ομιλητές ε, έθιξαν ζητήματα ανθρωπινών δικαιωμάτων και εξέφρασαν ανησυχίες. Έχουμε κατεπίγουσα λοιπόν την ε, ανάγκη να αντιμετωπιστούν ζητήματα επιτήρησης ε, τα οποία μάλιστα προξενούν και τριβές μεταξύ κρατών μελών και ημών και των διατλαντικών εταίρων μας. Ε, νομίζετε ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και εάν ναι, πώς μπορούμε να περιλάβουμε ακόμη και να ενσωματώσουμε σε μια τέτοια νομοθεσία το ζήτημα των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Επίσης, κρίσιμη σημασία μου φάνηκαν αυτά που είπε ο κύριος ο καθηγητής Στιούαρτ για την προσέγγιση της αλυσίδα προμηθειών και εγώ μιλώντας πάλι από την ε, οπτική του εμπορίου ε, μπορώ να πω ότι δεν μιλάμε πλέον στον κόσμο των εθνικών οικονομιών αλλά σε ένα κόσμο με παγκόσμιες αλυσίδες ε, προμηθειών και οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε πρέπει αυτό τον παράγοντα να τον λαμβάνουμε πάντα υπόψη. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε τώρα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τούνα Κέλαμ για να μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και στους τρεις ομιλητές, γιατί πραγματικά το να ε, μοιράζεστε μαζί μας ε, της γνώσης και την εμπειρογνωμοσύνη σας είχε πολύ μεγάλο νόημα σήμερα. Ήταν κάτι που χρειαζόμαστε και μας εμπλούτησε τις γνώσεις. Οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες, όπως είπατε, είναι μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο, όμως, ε, όπως είπατε, χρειάζονται βελτίωση, διότι τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν, τα ρί. Και η λέξη κλειδί είναι η ανάγκη αναθεώρησης του συστήματος. Αναφέρατε ότι Χρειάζεται να αναθεωρήσουμε τους ορισμούς, τα κριτήρια ελέγχου, τον ορισμό ε, των εξαγωγών, ε, τον κατάλογο, τη λίστα ε, ελέγχου. Το πρόβλημα με όλους αυτούς τους ορισμούς είναι ότι είναι αμφίσιμοι. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Δεύτερον, Έχω μια σειρά ερωτήσεις ε, σχετικά με τα παραδοσιακά προβλήματα συνεργασίας, συντονισμού, εφαρμογής, ε, διαφάνειας. Νομίζω ότι ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν έχει να κάνει με τα διάφορα επίπεδα εφαρμογής στα κράτη-μέλη, ειδικά τα μικρά κράτη-μέλη που έχουν περιορισμένες τεχνικές δυνατότητες έχουν πρόβλημα. Πολλά κράτη ε, δεν ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις τους να έχουν εσωτερικά συστήματα συμμόρφωσης. Τι μπορεί να γίνει με αυτό. Τέλος, πραγματικά με έχει ανησυχήσει το γεγονός ότι τα προγράμματα για την κατάρτιση και τη δημιουργία ικανονίτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν οικονομική βάση, όπως υπόθηκε. Και ένα πρακτικό ερώτημα τώρα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, απαιτείται να εφαρμόζουν εσωτερικά μέτρα και μηχανισμούς συμμόρφωσης για να συμμορφώνονται με τις ε, επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τεχνολογίες διπλής χρήσης. Υπάρχουν σήμερα επιπτώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών των διατάξεων. Πώς έχει το πράγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κέλαμ. Η κυρία Λέζινγκ Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Μιλάω γερμανικά, δεν ξέρω αν θέλετε να βάλετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την, ε, την εμπειρογνωμοσύνη σας. Από τη δική μου πλευρά να πω εκ των προτέρων ότι υποστηρίζω την αξιολόγηση που εμείς έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κοινή θέση σχετικά με τον έλεγχο εξαγωγών των πλεισμών. Πολλά μπορούν βέβαια να βελτιωθούν για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και συμμερίζομαι την εκτίμηση ότι αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας με την τρισδιάστατη εκτύπωση και Πράγματα που ως τώρα δεν είχαμε καν σκεφτεί. Από την άλλη να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ απεσιόδοξοι Είμαι απεσιόδοξη μάλλον για το κατά πόσο υπάρχει πολιτική θέληση ε, ε, να βελτιωθεί αυτή η κοινή θέση και πραγματικά να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι εξαγωγών. Να δούμε λίγο ποια είναι τα συμφέροντα από την πλευρά των βουλευτών. Ίσως υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά στην ουσία αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ε, πόσο μεγάλη σημασία έχει να γίνει αυτή η βελτίωση. Στην τελευταία νομοθετική περίοδο έγραψα, ε, εκπώνησα μία έκθεση για αυτήν εδώ την Επιτροπή σχετικά με αυτά ακριβώς τα θέματα. Ε, είχα συγκεκριμένες αναφορές στην εμπειρογνωμοσύνη του Σύπρη και γενικά μιλούσα για τη βελτίωση της κοινή θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αυτή ε, έλαβε πολλές ε, ε, τροπολογίες από το ΕΛΚ και στην Επιτροπή καταφέρανε να περάσουν όλες αυτές τις ε, τροπολογίες, οπότε στο τέλος η έκθεση δεν ήταν πια δική μου και την καταψήφισαν όλοι, δηλαδή πήγε στα σκουπίδια. Γενικά, επειδή αυτή η πλευρά είναι πολύ ε, αριστερή θα έλεγα. Ε, Ήταν μάλλον πολύ αριστερή αυτή η τάση γιατί την έκθεση την είχαν πολύ εξάρει η Ευαγγελική Εκκλησία και ούτω καθεξής. Γενικά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική θέληση για την εφαρμογή, ε, γιατί οι τεχνικές και οι οικονομικές δυνατότητες θα πρέπει να βοηθήσουν σε καλύτερη ε, σε βελτίωση του εξοπλισμού, επίσης ε, στο να έχουμε μία καλύτερη θεματική κάλυψη στο επίπεδο της ασφάλειας, του ανταγωνισμού, ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν πολιτικά και δυστυχώς ως τώρα η δική σας εμπειρογνωμοσύνη δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους βουλευτές σε αυτό το κοινοβούλιο. Δεν την ακούν πραγματικά. Ευχαριστούμε την κυρία Λέζινγκ. Να πω, λέει η πρόεδρος, και αυτό ε, το απευθύνω και στους τρεις ε, συμμετέχοντες στο πάνελ, αλλά είναι και η προφανής αλήθεια ότι πραγματικά το περιβάλλον στην ασφάλεια αλλάζει όχι απλά γρήγορα, αλλάζει ταχύτατα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω. Κάποιοι από τους εμπειρογνώμονες μας λένε ότι στην ουσία γίνονται ριζοσπαστικές ε, αλλαγές εκ των βάθρων στον κόσμο που ζούμε. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε πολύ διαφορετικές απειλές και για την εδαφική κυριότητα των κρατών μας και στην επικράτεια μάλλον των κρατών μας, αλλά και στη γειτονιά μας. Έχουμε ήδη συνηθίσει στην ανάγκη για μια άμυνα κατά της τρομοκρατίας και έχουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση στα ανατολικά. Για πολλά κράτη-μέλη αυτό ήταν κάτι απροσδόκητο. Εμείς από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ε, το είχαμε ήδη δει. Η ρωσική πολιτική, τουλάχιστον από το 2007 και μετά, ήταν ε, προφανής. Το ερώτημά μου είναι, εάν το να ληφθεί υπόψη ο, ο έλεγχος ε, των προϊόντων διπλής χρήσης, στην ουσία σημαίνει να παρατηρούμε και αυτά τα φαινόμενα. Ξέρω ότι ο πόλεμος της προπαγάνδας είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη, όχι μόνο του ΝΑΤΟ, μετά τη δημιουργία του κέντρου αριστείας του ΝΑΤΟ που είναι ακριβώς ε, επικεντρωμένο στις στρατηγικές ε, επικοινωνίες και έχει την έδρα του στη Ρήγα, αλλά και μετά από πολλές ε, ανακοινώσεις της Φερντερίκα Μοκερίνη, της είπα της εκπροσώπου, Ε, που στην ουσία ε, έκαναν πολλές ε, μονάδες και της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να μπουν σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει κάποια λογική πίσω από τον τρόπο που σκεφτόμαστε για αυτές τις απειλές και πραγματικά τι μέτρα νομίζω, τι μέτρα λαμβάνονται για τον έλεγχο προϊόντων διπλής χρήσης κατά τη διάρκεια μάλιστα της ε, ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το διάστημα. Το τρίτο επίσης, η TTIP, η Διατλαντική Συμφωνία, η οποία έχει πρόβλεψη, ε, που δεν έχει πρόβλεψη για την ε, άμυνα. Υπάρχει κάποια προσπάθεια ενοποίησης ή έστω προσέγγισης των καθεστώτων για τους ε, ελέγχους εξαγωγών προϊόντων διπλής χρήσης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών εταίρων. Σίγουρα όλοι προσπαθούμε να βγούμε από την οικονομική κρίση. και το κομμάτι του ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ξέρουμε ότι για να διατηρηθούν οι αμυντικές βιομηχανίες, χρειαζόμαστε αυτά τα προϊόντα διπλής χρήσης. Χρειαζόμαστε αυτό το κλάδο. Από την άλλη πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις προκλήσεις και τις άμεσες απειλές ε, στην ασφαλειά μας. Αυτά πώς τα εξισορροπείτε. Τώρα, με την ίδια σειρά θα ζητήσω από τα μέλη του πάνελ να δώσουν τις απαντήσεις τους και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Βίνκλερ για να καθοδηγήσει τη συζήτηση. Ο κύριος Κατσότη έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που διατυπώσατε. Καταρχάς, η ανάγκη για μια πιο συνεκτική προσέγγιση. Ο κύριος Βίνκλερ αναφέρθηκε σε αυτή. Σαφώς και χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά εδώ Θα ήθελα να σταθώ στην ιδιαιτερότητα που ξεκίνησε, που ανέφερα στην αρχή της παρουσίασής μου. Έχουμε θέματα εθνικής ασφαλείας, έχουμε θέματα διεθνούς εμπορίου και όπως πολύ σωστά είπατε, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ των τομέων αυτών και ορισμένες φορές η πρόκληση είναι να βρούμε την κατάλληλη προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος ε, δεν αναφερόμαστε μόνο στην διπλή χρήση, διότι η διπλή χρήση είναι μία από τις πτυχές ε, και είναι και ένα μέσο που θα μπορούσαμε να αλλάξουμε και να χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε συγκεκριμένους ελέγχους στον κανονισμό για να μην έχουμε και παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν όμως ε, και κάποια άλλα μέσα στη διάθεσή μας βεβαίως. Υπάρχουν κυρώσεις, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί για κάποιες ε, ε, πτυχές, για το βασανισμό π.χ. και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά έχουν ε, στοιχεία οικονομικά, εμπορίου, ασφάλειας και πολιτικά στοιχεία και όλα αυτά τα εξετάζουμε από κοινού. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ε, Για να μείνω στον ίδιο τομέα, η κυρία Φωτίγκα αναφέρθηκε σε μια αναπάντηχη απειλή και ε, τη δυνατότητα ε, υπάρχουν στην Ανατολή. Η Ρωσία είναι τμήμα ε, μέλος του Άρσενα και συμμετέχει στις συζητήσεις, αλλά στις κυρώσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις για προϊόντα διπλής χρήσης και έχουμε και αντιμετωπίσει κάποια από αυτά τα θέματα. Βέβαια θα πρέπει και εδώ να είμαστε προσεκτικοί να μην ε, κάνουμε κάτι το οποίο ε, μπορεί να φανεί εξ αρχής αποτελεσματικό και να δημιουργήσει προβλήματα στα άλλα μας θέματα. Για την TTIP ε, συζητάτε το ζήτημα. Βέβαια δεν αναμένουμε σύγκληση των δύο συστημάτων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν το σύστημά τους, αλλά ο διάλογος που γίνεται και ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε εθνικό επίπεδο ε, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία αυτά. Προσπαθούμε να υπάρχει μία σύγκληση σε στόχους τουλάχιστον όσον αφορά τη διαφορετική εφαρμογή από πλευράς κρατών μελών στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος από το King's College και ο κύριος Κέιλεμ. θα σταθώ σε κάτι που πολύ σωστά είπε η Σιμπίλ. Για τα διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής και αυτή η διαφοροποίηση στόχο έχουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Και αυτό μπορεί να είναι και κάτι θετικό. Υπάρχουν κάποιες περιοχές τις οποίες δεν υπάρχει ε, βιομηχανία προϊόντων διπλής χρήσης ή υπάρχει ελάχιστη πύρα από αυτόν και υπάρχουν και άλλες περιοχές στις οποίες ε, ο, η βιομηχανία συμμετέχει ε, ιδιαίτερα σε εξαγωγή τέτοιων προϊόντων και επομένως αυτό που έχει σημασία είναι να μην ε, υποσκάψουμε σε καμία περίπτωση την ασφάλεια, να μην δημιουργήσουμε παραθυράκια και να μην υποσκάψουμε και τη δυνατότητα ε, που μπορεί να έχει ένας εξαγωγίας εις βάρος κάποιου άλλου. Υπάρχει περιθώριο να βελτιώσουμε τα πράγματα, προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φυσικά υπάρχουν περιθώρια να γίνουν πολλά. Υπάρχει και αυτό το inner reach, η λύση σε εσωτερικό επίπεδο, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος προπολογισμό. Βέβαια, εδώ, ε, όπως γνωρίζουμε, ο προπολογισμό εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι που σα αποσχολεί. Είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να έχουμε κάποια πρόοδο. Εγώ στο παρελθόν ασχολήθηκα με τελωνιακά ζητήματα και θυμάμαι ότι όταν ε, ε συστήθηκε στην αρχή η ενιαία αγορά είχαμε μεγάλα σεμινάρια, ανταλλαγές ε, ανθρώπων που πήγαιναν ε, στα τελωνία άλλων χωρών να συνεργαστούν, κατάρτιση. Επομένως υπάρχει περιθώριο να βελτιώσουμε τα πράγματα και θα πρέπει να τα εξετάσουμε και από αυτή τη σκοπιά. Υπάρχει και μία ερώτηση η οποία τέθη για τα προγράμματα εσωτερική συμμόρφωσης, το ICP. Αυτά τα προγράμματα παρέχουν ε, σε κάποια κράτη-μέλη τη δυνατότητα πρόσβαση σε αδειοδότηση και αν δεν υπάρχει βεβαίω αυτό το πρόγραμμα δεν θα μπορεί κάποιο να έχει ε, άδεια αλλά το εξετάζουμε αυτό. Υπάρχει και μια ομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολείται με το θέμα αυτό. Προς το παρόν όμως δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Ε, υπάρξει παραβίαση, δεν υπάρχουν κυρώσει, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην εθνική νομοθεσία μπορεί να υπάρχουν τέτοιε προβλέψεις. Και θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να το εξετάσουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Μία τελευταία παρατήρηση για την TTIP. Βέβαια αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης, αλλά το συζητούμε γενικώ. Υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά κυρίως Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί κινούνται προς ε, μια πιο ανοιχτή προσέγγιση αδειοδότησης για να μειώσουν τους κινδύνους. Δυστυχώς ε, δεν αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Ε, έχουμε συνομιλήσει με τους Αμερικανούς επί του ζητήματος αυτού και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέλη των διαφόρων καθεστώτων. Και εδώ ε, υπάρχουν και όλες οι προκλήσεις αυτών που προσπαθούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για κάτι το οποίο ξεκίνησε σε εθνικό επίπεδο και τώρα που περνάμε σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ελλείψεις που έχουμε στον τομέα. Δεν θα συμβεί βέβαια αυτό εν μία νυχτή, θα χρειαστεί χρόνο και κόπο, αλλά ε, σίγουρα και προπολογισμό και υποστήριξη. Αυτά σας ευχαριστώ. Is this working? Yes. Λειτουργεί. Ναι, ο κύριος Στιουαρτ, παρακαλώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Θα ήθελα οι απαντήσεις μου να είναι σε ομάδες, γιατί υπάρχουν κάποια κοινά ζητήματα μεταξύ των σχολείων και των ερωτήσεων, αλλά και κοινέ λύσεις. Οπότε θα μιλήσω για τα τεχνικά ζητήματα από τη μία και τα πολιτικά από την άλλη. Τα τεχνικά είναι κάτι πέρα από την τεχνολογία. Ας αρχίσουμε λοιπόν με την πολιτική βούληση. Έχουμε εδώ ζητήματα ε, μεγάλης προβολής. αυτά τα ζητήματα ή έχουν να κάνουν με τη μεταφορά τεχνολογιών ε, παρακολούθησης, ε, ας πούμε, για την Αραβική Άνοιξη τέθηκε αυτό το ζήτημα. Μιλάμε για κυρώσεις στο Ιράν και διάφορα ε, θέματα προμηθειών. Όλα αυτά είναι υψηλής προβολής θέματα. Το να αναγνωρίσουμε κάτι τέτοιο και να δούμε πώς οι έλεγχοι επηρεάζουν αυτά τα ζητήματα στην ουσία μας κάνει να κατανοήσουμε και γιατί εφαρμόζονται όπως εφαρμόζονται οι έλεγχοι και γιατί δίνεται τόση έμφαση. Ο κανονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατά κάποιο τρόπο στατικός. Ναι, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδώσει τη λίστα, αλλά αυτό έρχεται από τους ε, ελεγκτές κυρίως. Τώρα για τη δυνατότητα αντίδρασης, ε, ε, να πω ότι είναι κάτι καλό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά θα έπρεπε να σκέφτεται για τις εξελισσόμενες ε, προκλήσεις στην ασφάλεια και για πώς αυτό θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει μέσα από τους ελέγχους και μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτό το θέμα και στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν υπήρξε πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει από την Κομισιόν, από το GRC γενικά μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Υπάρχει μια κατάρτιση η οποία πάει καλά, μπορούμε να την συνεχίσουμε. Τεχνικές αξιολογήσεις, αναφέρθηκε πολλές φορές η τρισδιάστατη εκτύπωση. Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι και απεσιόδοξος, αλλά έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, ε, εμείς στο Kings ε, προσπαθούμε να εξετάσουμε αυτές τις τεχνολογίες και να δούμε πώς πάνε. Να πω λοιπόν ότι αυτές οι τεχνολογίες ε, στην ουσία εξελίσσονται γρήγορα, όμως αυτές που έρχονται ως, στο άμεσο μέλλον δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση το πλαίσιο των ελέγχων. Επίσης, για την καθοδήγηση. Μιλάω και πάλι για τον ε, κανονισμό, για τις κανονισμούς και τα προγράμματα εσωτερικής συμμόρφωσης των εταιριών. Έχω αφιερώσει πολύ χρόνο σε αυτά τα θέματα, στον τομέα των οικονομικών και των ε, μεταφορών. Έχω αναφέρει την ακαδημαϊκή καθοδήγηση που έχει πρόσφατα εκδώσει το King's College ειδικά για τον τομέα των θαλάσσιων ζητημάτων. Και να πω ότι πάμε πέρα από τους κανονισμούς. Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν χρειάζεται περαιτέρω καθοδήγηση, η οποία βέβαια δεν είναι νομικά δεσμευτική, αλλά καλύπτει ένα κενό. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν υπήρχε κάποια τέτοια περίπτωση, ποιος θα ήταν ουσιαστικά υπεύθυνο ως άνθρωπο γι' αυτό. Επίσης ε, συζητήθηκε η δυνατότητα τεχνικής αντίδρασης ε, στην ανακοίνωση. Θα βοηθούσε λοιπόν ε, να ασχοληθούμε με πολλά από αυτά τα σημεία για να λύσουμε το ζήτημα. Λοιπόν, τώρα, για το τι γίνεται όταν υπάρχουν παραβιάσεις. Δεν νομίζω ότι γίνονται και πολλά ή δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός μηχανισμός παρακολούθησης των παραβιώσεων. Το να πάρει κανείς στοιχεία από την κοινωνία των πληροφοριών, βέβαια, που κάνουμε στο King's College, είναι κάτι που βοηθάει. Γιατί παίρνουμε μια εικόνα προς τα που πάντα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών ε, είναι κάτι που πρέπει να γίνει και σε αυτό το τομέα πραγματικά χρειάζεται. Δίνω το λόγο στη συνάδελφο τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Μπάουρ. Ευχαριστώ. Πολύ καλές ερωτήσεις. Οι προλαλήσαντες κάλυψαν, κάλυψαν μεγάλο φάσμα θεμάτων. Το θέμα, το ερώτημα το σχετικό με την ολοκληρωμένη προσέγγιση καταρχάς έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει τα πάντα να ενταχθούν στο ίδιο μέσον. Ε, δεν θα έχει καιρό, ε, μάλιστα. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να ε, υπάρχει επαρκής ροή πληροφοριών και συντονισμός μεταξύ των διαφόρων φορέων. Και επίσης Υπάρχουν ζητήματα τα οποία προσκρούν σε διαφορετική ε, σε κατακαιρματισμένη προσέγγιση, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές ομάδες ατόμων που ασχολούνται με διαφορετικά ζητήματα, με διαφορετική θεώρηση ενδεχομένως, καλή γνώση των θεμάτων, αλλά που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στο, χώρο, στο επίπεδο εργασίας πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα ε, νομοθετήματα τα εφαρμόσουν διαφορετικοί άνθρωποι, λένε πάντα τα ίδια νομοθετήματα. Το ίδιο αφαιρεπεί να το δούμε σαν εισαγωγές ή εξαγωγές όπλων που ρυθμίζουν και ελέγχουν τα, μάλλον που ελέγχουν τα τελωνία. Ζητήματα υπήρχαν επίσης προς την ε, κυβερνοεπιτήρηση. Ξέρω ότι υπάρχει και μια προηγούμενη ακρόαση στο θέμα αυτό που έχετε κάνει. Ε, ναι, έχουμε ιδιαίτερα υπογραμμίσει την πτυχή των ανθρωπών δικαιωμάτων, της ασφάλειας. Υπάρχει όμως και η άλλη πτυχή, που επίσης αναφέρεται σε μια ανακοίνωση που είναι οι συνέπειε για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ολόκληρο κάνιστρο λοιπόν ζητημάτων που δίνει και πολλές δυνατότητες για προκλήσεις, για επιθέσεις κατά κρίσιμης σημασίας υποδομών κτλ. Όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν. Έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση, μάλλον δεν έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση, αρχίζει μόνο. Και οι τεχνολογίες εποπτείας ή επιτήρησης έχουν ενταχθεί τώρα πλέον στον κατάλογο, αλλά δεν κλείνει με αυτό η υπόθεση. Υπάρχουν διαφορετικοί και αμφίσιμοι ορισμοί. Οι ορισμοί βεβαίως πάντα προσφέρουν ένα πεδίο ερμηνείας και αυτό ισχύει οπωσδήποτε για τα ευρωπαϊκά προϊόντα διπλής χρήσης. Ένα παράδειγμα είναι ο κατάλογος ελέγχου. Εάν ένα σημείο, εάν ένα ε, αντικείμενο προϊόν απαιτεί έλεγχο σε ένα κράτος ε, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτεί άδεια, τότε θα πρέπει ο παραγωγός και σε άλλο κράτος να ζητεί την αντίστοιχη άδεια. Αυτό είναι η τερμηνίας όμως που θα πρέπει να αντιμετωπιστώ. για την μεταφορά ILO προϊόντος ε, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το ζήτημα δεν είναι το πρόγραμμα προσαρμογής, μάλλον τήρησης να είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά να υπάρχουν ποικιλία εργαλείων και οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμμορφώνονται με το πρόγραμμα συμμόρφωσης που ε, αρμόζει στα στις ιδιαιτερότητε και τα μεγέθη του, του καθενός. Δεν μπορεί ο μικρομεσαίο παραγωγός να έχει τα ίδια μεγέθη και κριτήρια συμμόρφωσης με τον επιστήμονα ερευνητή ή με τον μεγαλομεταφορέα. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα καλύψει ο σχετικό κανονισμό διπλή χρήσης και στα θέματα των αδικημάτων και διώξεων που με έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα στην ερευνητική μου σταδιοδρομία. Ε, και ναι μεν ε, πρέπει καταρχήν να δημοσιοποιούνται τα, οι ετοιμιγορίες των δικασταρίων αλλά δεν είναι εύκολο να βρει κανείς, να κάνει την αναζήτηση κανείς γιατί είναι πάντα περίπλοκη και η ορολογία που χρησιμοποιείται ε, και έτσι είναι δύσκολο να κάνει κανείς την έρευνα για να καταλήξει στις σχετικές αποφάσεις. Αυτό δυσκολεύει πολύ τα πράγματα και άρα για το ίδιο αδίκημα μπορεί κανείς, για τον ίδιο τύπο αδικήματος μπορεί στη Γερμανία να φυλακίσετε κανείς για 15 χρόνια, ενώ σε μια άλλη χώρα μπορεί να επιβάλλεται απλή ποινή φυλάξης 2-3 ετών ή μόνο χρηματικό πρόστιμο. Ε, αυτά λοιπόν είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δυναμικό Επίσης, είναι οι περιορισμοί δηλαδή με τους οποίους έχουν να κάνουν ανακριτές και δικαστικοί. Ένα άλλο ζήτημα Σαλωστομέας με συναφή πολλά ζητήματα, έχει να κάνει με το έλεγχο των εξαγωγών που θα πρέπει να προσδιοριστεί κατά τρόπον ώστε τα εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τεχνολογικά εκείνα προγράμματα που μπορεί να έχουν κάποιες, ε, κάποιο αντίκτυπο στην ασφάλεια και την τεχνολογία να καλυφθούν και από τον κανονισμό διπλής κρίσης αλλά και από μια σειρά ε, άλλων γενικών διευθύνσεων θα πρέπει λοιπόν και αυτό να καλυφθεί. Πολλά από τα προϊόντα όμως πάντα υπάγονται στον έλεγχο υπό τον κανονισμό διπλής χρήσης. Ας σταματήσω εδώ προς το παρόν για να ακούσω και άλλες ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο σε κάτι που είπε ο κύριος Γκαρτσότη για η ε, Ρωσία που συμμετέχει στο συγκεκριμένο καθεστώς, ακόμα και αν το λάβουμε αυτό υπέψη, εχθές ε, ακούσαμε την παρουσίαση της έκθεσης που ξεκίνησε ο Λέιτ Μπορίς Μιντσόφ και μετά την ε, συνέχισαν οι συνεργάτες του και παρουσίασαν ένα πολύ προηγμένο σύστημα και αυτό το σύστημα δεν ήταν θέμα ρωσικής εμπειρογνωμοσύνης και έπεσε στα χέρια φιλορωσικών επαναστατών ε, στην Ουκρανία πρόκειται σαφώς για παραβίαση των συμφωνιών του Μίνσκ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συζητήσουμε όσον αφορά ε, το κατά πόσο θα πρέπει να περιλαμβάνει σε κάποιο κατάλογο και ούτω καθεξής. Το ερώτημά μου αφορούσε ε, κυρίως τη δική μας την οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή και και την ε, πιέση μας προς τις συνδεδεμένες χώρες και χώρες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο συγκεκριμένα την Ουκρανία σε αυτή την περίπτωση. Η συνεργασία ε, σε πολύ προηγμένα προγράμματα, παραδείγματος χάρη, τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα, διότι υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά το πώς διαχειρίζονται τα ε, προγράμματα του κοινού εναόριου χώρου και του κοινού διαστήματος ε, και τι γίνεται με τα προϊόντα διπλής χρήσης εκεί. Αυτή ήταν η φύση της ερώτησής μου. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι είναι πολιτική η φύση των παρατηρήσεων και των ερωτήσεών μου. Ωστόσο, η συζήτηση αυτή έχει πολιτικοποιηθεί ιδιαίτερα. συζητούμε ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολύ ε, σημαντική ανάγκη για ασφάλεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ευρωπαϊκών λαών, των γειτόνων μας και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βίνκλερ για να συνεχίσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Επομένως, ε, θα ήθελα να στραφώ προς τους ε, προσκεκλημένους μας, τους εκπροσώπους των διαφόρων ενδιαφερομένων ομάδων. Βέβαια, δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε πολλές ερωτήσεις, πολύ περιορισμένο αριθμό λόγω της ώρας και θα ήθελα ε, όποιο παίρνει το λόγο να μας συστήνεται και από εκεί και πέρα να μας διατυπώνει την ερώτησή του και να είναι και πολύ συγκεκριμένο να λέει σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση από τους τρει ομιλητέ μας. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Ακά Φούνερ. Ε, εργάζομαι για την Ομοσπονδία Γερμανικών Εταιριών. Σας ευχαριστώ για το εργαστήριο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εμείς ε, οι Γερμανοί ε, πραγματικά αντιμετωπίζουμε το θέμα με μεγάλη σοβαρότητα όσον αφορά γενικά τις εξαγωγές των ευρωπαϊκών προϊόντων. Φυσικά το θέμα είναι ευαίσθητο πραγματικά να εξάρω τις εισαγωγικές παρατηρήσεις του κυρίου Βίνκλερ, ο οποίος ε, αναφέρθηκε στο θέμα και επειδή δεν υπάρχουν πολλοί βουλευτές εδώ, θα ήθελα να ζητήσω από τη Γραμματεία να δώσει τις παρουσιάσεις σε όλους τους βουλευτές. Ευχαριστούμε τον κύριο Φορούγκελν. Κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Δεν βλέπω κανέναν να σηκώνει το χέρι του. Ah, excuse me, please. Hi. Um... <clears throat> Γεια σας. Ονομάζομαι Μάινες Νεριούς. Είμαι ε, εδώ εκ μέρους της ψηφι... βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτό το εργαστήριο. Θα ήθελα να τονίσω κάποια από τα ζητήματα εκ μέρους ε, της ψηφιακής Ευρώπης, ε, γιατί εκπρόσωπούμε την ε, ICT, την IT και τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες για τους καταναλωτές. Υπάρχει παντού σχεδόν κρυπτογράφηση στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής για να προστατευτούν οι χρήστες και οι καταναλωτές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν για τα δεδομένα και το παλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της διπλής χρήσης, γιατί ένα αντικείμενο διπλής χρήσης μπορεί να αποτελεί απλώς ένα μικρό γρανάζι μιας βρύτερης μηχανής, αλλά πραγματικά θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν δεδομένα που μπορεί να αφορούν στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που έχουν αυτά τα στοιχεία, καθώς μια ολόκληρη εταιρεία μπορεί να επηρεάζεται από ένα τέτοιο αντικείμενο ή ολόκληρες οι εξαγωγές τους. Ίσως επίσης θα πρέπει να απαλλαγούμε από ελέγχους σε κάποια χαμηλής ε, ε, σημασίας προϊόντα, ας πούμε, ημιαγωγούς. Ε, το αμερικανικό σύστημα ε, ελέγχου εξαγωγών έχει κάποια τέτοια διάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω αν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής νέων γενικών αδειών δεδομένων των προκλήσεων που είχαμε στο παρελθόν. Αυτές τις ερωτήσεις έχω. Ευχαριστώ. Και άλλη μια ερώτηση, παρακαλώ έχετε το λόγο. Είμαι από το κελτικό, α, κελτική βιομηχανία. Έχω, μια, ε, έχω δύο ερωτήσεις. Ο κύριος Γκαζότη ανέφερθηκε με τη λέξη ευρωπαϊκός στους, ε, στα Μητρώα. Ε, τι ακριβώς εννοούσε με τα Μητρώα μετά για ε, τον κύριο από το Ζήπρη. Πώς πρέπει να ρυθμίζεται η τεχνολογία των πληροφοριών, τα άειλα προϊόντα, όπως ας πούμε το λογισμικό, είναι κάτι από αυτά που στην ουσία, διαγράψ... Ε, στην ουσία μας ε, διαγράψετε με την ομιλία σας και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χόρκατ. Έχουμε μια σειρά ερωτήσεων, οπότε δίνω το λόγο στα μέλη του πάνελ και θα ήθελα να ορίσετε αν ε, πραγματικά μπορούμε να δημοσιεύσουμε τις παραδοσιάσεις σας όπως ζητήθηκε. Έχετε το λόγο. Thank you. Ε, σας ευχαριστώ για τις δύο ερωτήσεις που αφορούσαν τη δική μου παρουσίαση. Ο έλεγχος ορισμένων προϊόντων. βασίστησε σε ένα κατάλογο τον οποίο προσδιορίζει αρκετά επακριβώς έως και πολύ επακριβώς ο κανονισμός. Δηλαδή μόνο αυτά που ορίζει το καθεστώς μπορούμε να περιλάβουμε στον κατάλογο ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα προϊόντα. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει κάποια αλλαγή στο μέλλον. Προ το παρόν η πρόταση επιτροπή ορίζεται από την εντολή που τη χορηγεί ο κανονισμό. Αλλαγή δεν υπάρχει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμβάλλουμε στο καθεστώς στο να γίνονται έλεγχοι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, οργανώνουμε δηλαδή όσο περισσότερο γίνεται τη συμβολή στο σύστημα αυτό των κρατών μελών. Βέβαια, γιατί βασικά αυτό μπορώ να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλος, ενώ είναι η Ρωσία. Το σημειώνω αυτό. Και βέβαια είναι και επιμέρους κράτη-μέλη αλλά όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Για την κρυπτογράφηση και τους ελέγχους. Έχουν ήδη ε, συστήματα αδειοδότησης ορισμένα κρατημέλη. Στην αξιολόγησή μας παρακολουθούμε και διερευνούμε την ιδέα ενδεχόμενης αδειοδότησης πανευρωπαϊκής που να καλύπτει και ζητήματα κρυπτογράφησης. Μέχρι και έχουμε φτάσει. Για την έρευνα. Με την Παύλα εκεί πέρα. Γιατί δεν ήταν παρένθεση νομίζω. Υπάρχουν γνώσεις και τεχνογνωσία και τεχνολογία και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε την, τον κίνδυνο να καταλήξουν σε χέρια ακατάλληλα. Ένα θέμα πολύ λεπτό, όσο και σοβαρό. Γιατί εδώ μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τη θεώρηση ευατηρίου για επιστημονική έρευνα σε κάποιον που περνάει τα σύνορα με λάθος ιδέες στο κεφάλι. Θα τον σταματήσουμε. Μπαίνει αυτό στον ελέγχο διπλής χρήσης. Αυτή είναι νομίζω μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις που έχουμε. Και όπως είπα, έχει τεράστια σημασία η ε, ανταλλαγή πληροφοριών, η κατανομή των, το μοίρασμα των πληροφοριών. Ευχαριστώ για να απαντήσω κι εγώ. στο ερώτημα για την κρυπτογράφηση. Έχω περάσει χρόνο πολύ με καταλόγους ελέγχου, κρυπτολόγηση, επιχειρήσεις κτλ. Εμένα αυτό το ζήτημα της κρυπτολόγησης δεν είναι το ε, αγαπημένο μου θα έλεγα. Στην υπόθεση αυτή δεν θέλω τόσο πολύ να το αγγίξω. Γιατί όταν συζητούμε με επιχειρήσεις και τους ρωτούμε τις, ε, τους κινδύνους ε, από την τεχνολογία, Πολλά, πολύ συχνά μας λένε ότι δεν είναι κρυπτογράφηση το πρόβλημα όσο το προϊόν μέσα στο οποίο είναι ενσωματωμένοι. Και αυτό συνεπάγεται χαμηλό ποσοστό άρνησης ελέγχου λόγω κρυπτογράφησης. Άρα υπάρχουν δυνατότητες να ξαναδούμε το θέμα της κρυπτογράφησης. Υπάρχουν τρόποι να το επιτύχουμε φαίνεται ότι υπάρχει μία πρόταση για αναδιατύπωση κειμένου. Ίσως και ελπίζω τα θέματα των εμπορικών εξυπηρετητών σερβερ να βγουν από τον έλεγχο προϊόντων και εν ολίγης νομίζω ότι το καλύτερο είναι να βρεθεί η πιο ισορροπημένη λύση ώστε να εξασφαλίσετε ένας αποτελεσματικός έλεγχος. Thank you. I'd like Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις για τον έλεγχο του λογισμικού. Δεν νομίζω ότι ο έλεγχος του λογισμικού στον κανονισμό ε, για τη διπλή χρήση είναι ο, ο απαραίτητος, αλλά είναι λογικός. Θέλουμε να έχουμε καλό λογισμικό και τεχνολογία ε, και ελέγχουμε κάποια αντικείμενα γιατί έχουν κάποιες δυνητικές εφαρμογές, ε, ε, προγράμματα βιολογικών, πυρηνικών, χημικών όπλων και έχουν και διαφορετικές εφαρμογές από τα συμβατικά όπλα. Αυτή είναι η συζήτηση και από εκεί και πέρα συζητώνται πιθανές χρήσεις τεχνολογίας κυβερνοεπιτήρησης. Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι μάλλον ξεχωριστό. Αυτό το οποίο ε, είναι μια σημαντική διαφοροποίηση είναι τι γίνεται όταν ελέγχουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν και ότι έχει χρήσεις για παράδειγμα σε προγράμματα πυρηνικών όπλων και δεν ελέγχουμε μόνο το αντικείμενο αυτό καθευτό αλλά και το σχετικό λογισμικό και τη τεχνολογία. Παραδείγματο χάρη, τρισδιάστατες εκτυπώσει στο μέλλον, όπως ανέφερε και ένα συνάδελφο, ε, ο οποίος είναι ειδήμων σε θέματα βιολογικά, στο μέλλον θα μπορούμε να έχουμε ε, δυνατότητα να τυπώνουμε με τρισδιάστατο εκτυπωτή ε, πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να διανοηθούμε καν. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ποιο είναι ο σκοπός των ελέγχων, πώ μπορούμε να του επιτύχουμε αποτελεσματικά μεν, αλλά ταυτόχρονα πώς μπορούμε να αποφύγουμε, όπως έλεγε και κάποιος προηγούμενος ομιλητής, να ε, πιάνουμε πολλά αθώα ψάρια και τις μαρίδες, ενώ προσπαθούμε να πιάσουμε τα μεγάλα ψάρια. Και αυτή είναι και η μεγάλη δυσκολία με τους ελέγχους ε, προϊόντων διπλής χρήσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους ομιλητές, αυτούς τους οποίους έθεσαν τις ερωτήσεις. Ε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ εκ μέρους της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, διότι μας δώσετε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση και από πλευράς ε, Επιτροπής ε, Διεθνούς, Εμπορίου μια φράση. Ίσως δεν είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα, αλλά είναι ένα σημαντικό συμπέρασμα αυτής της συζήτησης για τους ελέγχους των εξαγωγών των προϊόντων διπλής χρήσης. Δεν πρέπει τα πάντα να γίνονται μέσω κανονισμού. Νομίζω ότι η χρήση ήπιας νομοθεσίας και κατευθυντηριών γραμμών και καθώς επίσης το να ληφθεί υπόψη ε, η άποψη των ενδιαφερομένων και να τους εκπαιδεύσουμε ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, κύριε Συμπρόεδρε. Εκ μέρους της ε, Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για αυτή την κοινή συνεδρίαση. Να ευχαριστήσω ευγενικά και τους ομιλητές μας τρεις εξαιρετικούς ομιλητές για την πολύ σημαντική συνεισφορά τους και τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτήματά μας να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και τους εκπροσώπους του ακαδημαϊκού κλάδου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, του κλάδου και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι το απόγευμα η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 3 ακριβώς Πρόκειται για μία ακόμα κοινή συνεδρίαση. Θα συμμετέχουν και οι επιτροπές ε, Ήτρε και Ίμκο για ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Μπινκόφσκα. Παρακαλώ λοιπόν για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ.